Um, Θα ξεκινήσουμε. Έχω κάποιες ανακοινώσεις ως συνήθως. Η έκθεση της EIB, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου, όπως φαίνεται στην τελευταία ημερήσια διάταξη. Περνάμε τώρα στις ανακοινώσεις της Προεδρίας για την κατάσταση στους τριμερείς διαλόγους. Είχαμε ένα τέτοιο διάλογο για τις κεφαλουχικές απαιτήσει για θέματα ρευστότητας σκιωδών πιστοτικών δραστηριοτήτων κτλ και προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι τα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις συζητήσεις μέχρι το τέλος ε, του μήνα. Έχουν γίνει σε επίπεδο συντονιστών ορισμένες προτάσεις. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειες ε, και στα τρία θεσμικά όργανα σε επίπεδο τεχνικό και η επόμενη συνάντηση τριμερούς ε, διαλόγου θα γίνει στο Στρασβούργο στις 23 ε, Οκτωβρίου. Περνάμε τώρα στο σημείο 5, ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και παρουσίαση της εκθέσεως από τον κύριο Μάουρο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα θα σας πω τα βασικά της έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να υπάρξει αύξηση του κεφαλαίου της. Γι' αυτό η απόφαση του Συμβουλίου τον μήνα Ιούνιο ήταν θετική. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταστήσουν την αύξηση του κεφαλαίου της τράπεζας λειτουργική το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό είναι απαραίτητο για να κρατήσει το τριεπλό α την απαραίτητη αξιολόγηση γιατί δυστυχώς οι επενδυτές δεν θεωρούν πολύ ελκυστικές τις μετοχές της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και οι περισσότεροι επενδυτές προέρχονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μπορέσει λοιπόν να λειτουργήσει σωστά και χρηματοδοτικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να δημιουργήσουμε νέα χρηματοπιστωτικά μέσα που να βασίζονται στο σωστό συνδυασμό των πόρων από τη μία του προϋπολογισμού της Ένωσης και από την υψηλή ε, δανειοδοτική δυνατότητα που θα έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η πιλωτική φάση αυτών των ομολόγων, των διαφθορτικών ή των καλύτερα project bonds ε, θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013 για να επιτρέψουμε την ανάπτυξη νέων μέσων, μεικτών, δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να κατανείμει σωστά τις αρμοδιότητες των δύο πλευρών να δίνει εγγυήσει για την απαιτούμενη ευελιξία και να μπορεί να τραβάει πόρους και από τον δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να αποφύγουμε υπερβολικές γραφειοκρατικές παρεμβάσεις για αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται τις μορφές χρηματοδότησης σε οποιαδήποτε φάση αυτής βρίσκονται. Θα πρέπει να διευκρινιστούν σωστά οι εκ των προτέρων στόχοι και οι εκ των υστέρων μορφές ελέγχου της διαδικασίας και θα πρέπει η ΕΕΠ να κρατήσει την δική της ανεξαρτησία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής και να χρησιμοποιήσει τους πόρους της με βιώσιμο τρόπο. Θα πρέπει επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δώσει εγγυήσεις περισσότερης διαφάνειας δίνοντας περισσότερα στοιχεία εκεί όπου γίνονται έλεγχοι για αυτούς οι οποίοι ωφελούνται και για τους ενδιαμέσους στις χώρες υποδοχής, αν θέλετε, των χρημάτων, των επενδύσεων. Πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα όχι πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά απουσίας μιας ίδιας διαχειριστικής ικανότητας από πλευράς αυτών που αποδέχονται τις παρεμβάσεις. Αυτό είναι επιβραδυντικό για την ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να, να συνεχίσει να, να συγκεντρώνει την προσοχή της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας επίσης και μέσα μικροχρηματοδότησης, συνεργαζόμενοι με πιστοτικά ιδρύματα που ειδικεύονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και τους λεγόμενους μη συμβατικούς πιστοτικούς ενδιαμέσους. Εμείς λοιπόν ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να στηρίξει και την κοινωνική οικονομία που δημιουργεί δυνατότητες ευημερίας και θέσεις εργασίας μέσω ειδικών μορφών δανειοδότησης και προγραμμάτων εγγυήσεων ε, μπορούμε να λάβουμε υπόψη καλύτερα και τις συνέργειες που υπάρχουν με τη λεγόμενη Social Business Initiative πρωτοβουλία κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν και νέες παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού, στον τομέα της δημιουργίας που έχει χτυπηθεί άσχημα από την χρηματοπιστωτική κρίση. Η Ευρωπαϊκή τράπεζα, αυτή η τράπεζα επενδυτική, πρέπει να λειτουργήσει, δυστυχώς για αυτήν αν θέλετε, σε τομείς όπου οι περικοπές από πλευράς του δημοσίου είναι οι υψηλότερες. Οι περικοπές γίνονται επίσης όχι μόνο από τις κυβερνήσεις αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα αυτό το δείχνει η συζήτηση που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον τελευταίο καιρό για το MFF έρευνα, καινοτομία, πολιτισμός, ενεργειακή αποδοτικότητα, συνέργειες με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ΚΑΠ, διαρθρωτικά ταμεία. Σε όλα αυτά λοιπόν πρέπει να υπάρξει μία πρόοδος. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες της Μεσογείου και οι υποψήφιες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλείται να χρηματοδοτήσει υποδομές και πάντα μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταπολεμήσει τις αρνητικές συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών και να υποστηρίξει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Και στα πλαίσια των εξωτερικών της δραστηριοτήτων θα πρέπει να κρατάει την κοινοτική της φύση θα έλεγα και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες μορφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεμβαίνοντας στις χώρες τις οποίες μπορεί να κάνει διαφορά όπως ακριβώς στις χώρες γειτονίας που εντάσσονται στην πολιτική γειτονίας σε χώρες οι οποίες την χάνουν συνεργασία στα πλαίσια των προγραμμάτων συνεργασίας και ανάπτυξης είναι Ευρωπαϊκή Τράπεζα και έχει ιδιαίτερο ρόλο να παίξει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις γειτονικές χώρες και στα πλαίσια της άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ τώρα να μπω σε λεπτομέρειες σε άλλα θέματα, αλλά κάποια μόνο σημεία θα πρέπει ίσως να θίξω. Πάντως, όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, έχουμε πρόβλημα, αν θέλετε, μεγέθους της παρουσίασης και γι' αυτό είμαι υποχρεωτικά συνθετικός και συνοπτικός. Περιμένω τις τροπολογίες σας που θα καταστήσουν το κείμενο ε, καλύτερο. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 25 η Οκτωβρίου. Είχα μια ανεπίσημη συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Από εκεί βγήκαν κοινέ απόψεις και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Okay, uh, Καλώς. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Κούτας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μάουρο για το ανοιχτό του πνεύμα και για την επιθυμία του να συνεργαστεί στενά με τους σκιώδεις. Αυτό φάνηκε από την συνάντηση που οργάνωσε ο ίδιος λίγο πριν. Το σχέδιο θα έλεγα ότι είναι καλά ισορροπημένο. Θέλω να αναφερθώ σε μερικά συγκεκριμένα στοιχεία που εγώ θα ζητήσω να προσθεθούν υπό τη μορφή τροπολογιών. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ζητήσουμε από την ΕΤΕ να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες περιφέρειες χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλής απασχόλησης με επενδυτικό έργο αλλά και με τα ομόλογα έργου. Τώρα για την μελλοντική τραπεζική ένωση πρέπει να δούμε τι ρόλο θέλουμε για την ΕΤΕ εκεί μέσα. Τρίτον, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να βασίζεται λιγότερο σε ενδιάμεσους, διότι πολλές φορές τα οικονομικά δεν φτάνουν τελικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά μένουν στους ενδιάμεσους. Μία λύση λοιπόν θα ήταν η Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων να χρησιμοποιήσει περισσότερες ε, risk sharing facilities. Θέλω επίσης να ζητήσω από τον εισηγητή να δεχτεί, αν θυμόσαστε, η Επιτροπή μας ζήτησε με τη γνωμοδότηση της πέρυσι ή να φτιάχνει τον ε, δικό της κατάλογο με τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες και νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στο αίτημά μας αυτό. Όπως είπε και ο εισηγητής, η διαφάνεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική πτυχή. Πιστεύω ότι πρέπει να ενημερώνετε το κοινό όχι μόνο για την επιλεξιμότητα και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αλλά και για τους ενδιάμεσους και για τους ε, δικαιούχους και για τα ποσά που αποφασίζονται κλπ. Υπάρχουν μερικά σημεία λοιπόν τα οποία θέλω έτσι να θίξω και το έκανα και κατά τα άλλα προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί με όλους τους συναδέρφους για το θέμα αυτό. σε ευχαριστούμε. Ε, παρακαλώ. Θόδωρο, ναι, δεν σε έβλεπα. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για μια έκθεση που πραγματικά είναι πολύ ισορροπημένη, αλλά και για το πνεύμα συνεργασίας που έχει επιδείξει μέχρι τώρα. Θέλω όμω και να συμπληρώσω λιγάκι στην ίδια βάση στην οποία μίλησε και ο προλαλή σα. Πιστεύω και εγώ ότι στην Ευρώπη υπάρχουν περιφέρειες όπου η ανεργία είναι πάνω από 25% σήμερα. Συνεπώ, έχουμε και την Ευρωζώνη που σε μερικές περιπτώσεις δεν λειτουργεί. Γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια από 250 μονάδες βάσης από ένα σημείο της Ευρωζώνης σε κάποιο άλλο. Συνεπώς, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δραστηριοποιηθεί στις περιφέρειες ακριβώς αυτές. Γιατί στην πραγματικότητα κανένας άλλος δεν θα το κάνει, αν δεν το κάνει εκείνη. Και είναι μεγάλη απώλεια να έχουμε το ένα τέταρτο του ενεργού πληθυσμού μιας χώρας ή το ένα πέμπτο στην ανεργία και να μην κάνουμε τίποτα απολύτως. Είναι μια τεράστια οικονομική αποτυχία αυτό. Πέρα από αυτό θέλω να υπογραμμίσω ότι ο τρόπος με τον οποίο τα ομόλογα έργου ετοιμάζονται σήμερα θα αποκλείσει αυτές τις περιφέρειες ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει επίσης να προσέξουμε. Τέλος, πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλη αυτή η επενδυτική δραστηριότητα που θα αρχίσει τώρα είναι 0,3 του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό ποσό, μια πολύ μικρή επενδυτική δραστηριότητα στην πραγματικότητα, που σίγουρα δεν είναι αρκετή για να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση. Για άλλη μια φορά πάντως ευχαριστώ τον κύριο Μάουρο. Ευχαριστώ άλλος, κανείς από τους πράσινους, μήπως είναι εδώ κανείς που θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ο κύριος, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω με τη σειρά μου στον κύριο Μάουρο, εκ μέρους των Πρασίνων, ότι συμμεριζόμαστε ειλικρινά την ανάλυση του όσον αφορά τον ρόλο και τη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Τράπεζα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σήμερα φαίνεται να παίρνει ακόμα περισσότερη σημασία, μια που αποτελεί το εργαλείο δυναμισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής λιτότητας που ζούμε. Κατά τη γνώμη μου, μάλιστα, αποτελεί και το στοιχείο κλειδί για το σύμφωνο σταθερότητας, που εμείς προτιμάμε να λέμε ε, ανάπτυξης, και συμπληρώνει τον κοινοτικό προπολογισμό. Συνεπώς, ναι στις νέες δυνατότητες για δάνεια από πλευράς της ΕΤΕ, ναι στο να στοχεύει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ναι στην αύξηση του κεφαλαίου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι στην επιθυμία για διαφάνεια σε διοικητικό, δημοσιονομικό επίπεδο, δίκησης κτλ. Αλλά όλα αυτά γιατί με τη σκοπό με τι προτεραιότητες. Οι πράσινοι λοιπόν θα υποβάλουν, έχουν ήδη υποβάλει κάποιες τροπολογίες στην έκθεσή σας κύριε Μάουρο, οι οποίες προσπαθούν ακριβώς να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της στήριξης αυτής στην καινοτομία, της στήριξης αυτής στην αποτελεσματικότητα των πόρων, της στήριξης αυτής στις στρατηγικής σημασίας υποδομές. Θέλουμε να στοχεύσουμε καλύτερα τις επενδύσεις της ΕΤΕ υπέρ μιας πιο οικολογικής οικονομίας, δηλαδή υπέρ της ενεργειακής απόδοσης, υπέρ των αναλλακτικών πηγών ενέργειας, υπέρ ε, μεταφορών πιο βιώσιμων, ε, γενικά υπέρ ό,τι βοηθάει την ε, οικολογική αλλαγή στην οικονομία μας. Εμείς με τις τροπολογίες μας θέλουμε στην έκθεσή σας να προσφέρουμε έναν καλύτερο, μια καλύτερη κατεύθυνση όσον αφορά τις επενδύσεις της ΕΤΕ, ώστε να έχουμε μια πηξίδα που θα μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο Ντέρκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μάουρο για το έργο του στο σχέδιο έκθεση. Έχει δίκιο λοιπόν ο κύριο Μάουρο όταν λέει ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι χρήσιμο. Στη χρηματοδότηση ε, της οικονομικής ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διασφαλίσει την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξουν ορισμένες επιμέρους ρυθμίσει. Θα καταθέσω τροπολογίες οι οποίες θα βοηθήσουν νομίζω να γίνει σωστότερη η έκθεση. coffee break, sorry. Με συγχωρείτε, αλλά έκανα ένα διάλειμμα για καφέ. Θέλω λοιπόν να εξηγήσω σύντομα αυτές τις αλλαγές τώρα. Δηλαδή καταρχήν θα ήθελα να εξετάσετε αν θα ήταν δυνατόν να ενισχύσει κανείς τα προγράμματα τα οποία υφίστανται σε συνεργασία με την ε, ε, ε, τράπεζα ότι τα προγράμματα που ήδη υφίστανται απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση τώρα. Πρόκειται για εταιρείε οι οποίες θα επηρεάσουν άμεσα και την οικονομική ανάκαμψη σε τοπικό επίπεδο δημιουργώντας θέσεις εργασίας και, να, και αν στηρίξουμε τα προγράμματα αυτά στηρίζουμε τους πολίτες γι' αυτό και θα ήθελα να τα, τους ενθαρρύνουμε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως έχει ε, ζητήσει ε, μία σειρά κατευθυντηρίων γραμμών και ε, εντωμεταξύ ε, χρειάζονται να υπάρχουν τραπεζικές δυνατότητες για, να, για δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η συμμετοχή στον κίνδυνο είναι ένα βασικό επιχείρημα, δηλαδή θα πρέπει οι τράπεζες να μπορούν να επιτρέπουν πρόσβαση ε, στην χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να καθίσουμε να αξιολογήσουμε πολύ λεπτομερώς τη βιωσιμότητα του νέου μέσου και να δούμε πώς θα επηρεάσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την συμμετοχή στην ανάληψη κινδύνων σε, ένα δεύτερο, σε μια δεύτερη φάση ενδεχομένως και καλό θα ήταν να καταρτιστούν καλά προγράμματα και να μην ξεκινήσουμε να σπαταλάμε ε, χρήματα σε αμφίβολα προγράμματα τα οποία έχουν ε, ε, περιορισμένη δυνατότητα απορροφήσεως και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το γνωρίζει. Τέλος για τον ορίζοντα 2020 για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις πράσινες τεχνολογίες και την ανακύκλωση και ε, ε, η έλλειψη ορισμένων πόρων όπως καθαρό πόσιμο νερό μας επηρεάζει όλους και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά ολόκληρο, ολόκληρη την Ιφίλιο η οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί από την πρόοδο στον τομέα της ανακυκλώσεως και να επηρεάσει θετικά το περιβάλλον. Ευχαριστώ κύριος Χουντής. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή μας και καταρχήν να επαναλάβω κάποιες ε, συμφωνίες μας για να έχει υπόψη του ότι έχει και τη συνένεση της δικής μας και τη στήριξη και της δικής μας ομάδας σε βασικά σημεία της έκθεσης. Ε, και θα επαναλάβω ότι έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, σε συνθήκες κρίσης, με την ανεργία να μεγαλώνει σε πολλές χώρες, το πρόβλημα της ανάπτυξης να είναι ζητούμενο η πραγματική σύγκληση και το θέμα της κοινωνικής συνοχής να αμφισβητείται έως να απομακρύνεται ως στόχο είναι λογικό και ενισχύουμε την σημασία που υπογραμμίζει και ο εισηγητής του ρόλου που μπορεί να παίξει και το ακόμα πιο ενισχυμένο ρόλο που μπορεί να παίξει η Τράπεζα Επενδύσεων παρά το μικρό κύκλο δραστηριοτήτων σε σχέση με το συνολικό ΑΕΠ όπως τόνισε προηγούμενος συνάδελφος. Υπάρχουν δηλαδή μεγαλύτερε προσδοκίες για πιο στοχευμένη ε, χρηματοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να τα λύσει μόνο η Τράπεζα Επενδύσεων αυτά τα ζητήματα. Σωστό αυτό, είμαστε σύμφωνοι. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι εδώ στο διάστημα που εξετάζουμε ε, η συμβολή της ε, τράπεζας ήταν ορισμένες φορές διστακτική και αργή και θα το σημειώσω, το σημείωσε ο εισηγητής μας και είναι ένα θέμα βεβαίως, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο πράγμα. Η αναζήτηση ή η προσπάθεια να εξασφαλίσει την υψηλότερη κεφαλαϊκή θέση με τα 3α πολλές φορές την κάνει διστακτική στο να ανοίξει την επενδυτική της δραστηριότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο κατάλληλη θέση ισορροπίας και αν θα μπορούσε από λιγότερο ισχυρή κεφαλαϊκή θέση να αναπτύξει μια μεγαλύτερη δραστηριότητα αφού όπως είπαμε και εδώ συμφωνούμε όλοι υπάρχει μεγάλη απέτηση. Είναι όμως ένα πρόβλημα, δεν το θεωρώ ότι είναι εύκολο, εξήγησε ο εισηγητής μας που οφείλεται αυτό διότι δεν θεωρούνται αξιόπιστες οι, από την πλευρά των επενδυτών οι, οι χρηματοδοτήσεις από την πλευρά της ε, ε Τράπεζας Επενδύσεων εφόσον δεν έχει τα 3α αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πρόβλημα που προφανώς την κάνει πιο διστακτική, πιο αργή και λιγότερο αποτελεσματική στις παρεμβάσεις που υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Ε, δεύτερο, είμαι, ε, υπογραμμίζω και εγώ ότι πρέπει οι στοχευμένα, στοχευμένα οι προτεραιότητες να κινηθούν στις χώρες που έχουν σήμερα τα μέγιστα προβλήματα ε, οικονομίας ε, λόγω της κρίσης και λόγω μνημονιακών πολιτικών θα προσέθετα εγώ από την εμπειρία της ε, χώρας μου. Το θέμα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλες τέτοιες δραστηριότητες πολλές φορές δεν κολλάει μόνο, σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις που σωστά τις επισημαίνει ο εισηγητής, κολλάει σε αντιφατικές πολιτικές, από τη μια μεριά μνημονιακές απαιτήσει και από την άλλη μεριά οι απαιτήσει να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Και εκεί η Τράπεζα Επενδύσεων βρίσκεται κάπου στη μέση αδρανούσα, όπως τουλάχιστον κατάλαβα από τη συζήτηση που είχαμε με τον Πρόεδρο στην προηγούμενη ακρόαση που οργάνωσε η Επιτροπή μας Τέλος, ε, υπογραμμίζω και εγώ την ανάγκη της διαφάνειας στα φορολογικά ζητήματα, τους αποδέκτες των δανείων, αν μπορεί ο έλεγχος να είναι πιο αυστηρός προκειμένου να αποφευχθούν οι παραπομπές σε φορολογικούς παραδείσους και άλλες πρακτικές όπως και σε άλλες περιπτώσεις έχω αναφέρει ενδομιλικές τιμολογήσεις και ούτω καθεξής. Με βάση αυτό λοιπόν ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο για τη δουλειά που έχει κάνει. Οι τροπολογίες θα κινηθούν στο πνεύμα αυτών των συμπληρώσεων που θεωρούμε σημαντικές για την έκθεσή μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Uh, thank you very much. Is there... Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς που θέλει να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα. εκπρόσωπος Τιαπή, μήπως. Δεν ξέρω, αν έχουμε λίγο χρόνο, αν νομίζετε. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μάουρο για την πράγματι ισορροπημένη εκθεσή του. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, πιστεύω. Επιτρέψτε μου να κάνω όμως μερικά σχόλια σε σχέση με αυτά που άκουσα εδώ στην αίθουσα. Όσον αφορά το ομόλογα έργου, Γνωρίζετε ότι η φάση αυτή μόλις έχει αρχίσει. Τον Ιούλιο μόλις εγκρίνατε τη σχετική ρύθμιση και άρχισε να ισχύει από τον Αύγουστο. Έχουμε μπει στο αυλάκι, ξεκινούμε τη δουλειά, αλλά βέβαια χρειάζεται χρόνο για να ετοιμάσουμε καλά σχέδια. Ελέγχουμε και εξετάζουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες, την επόμενη περίοδο. Τώρα η αύξηση του κεφαλαίου και πάνω σε αυτό δουλεύουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε πράγματι την ε, οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη γενικότερα. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι το Μάρτιο ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε αμέσως. Αυτό που κάνουμε είναι πράγματι υπέρ των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων είναι και η μεταρρύθμισή μας αυτή, το αντικείμενο δηλαδή της μεταρρύθμισής μας που εγκρίθηκε πέρυσι. Θέλουμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο και σε υπηρεσίες και έχει ετοιμαστεί ένα σχετικό τμήμα που δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, ναι, λαμβάνουμε υπόψη μας και τέτοιες πρωτοβουλίες. Ήδη με την ε, μικροπιστώσεις, με το πρόγραμμα αυτό για τις μικροπιστώσεις, έχουμε ήδη ξεκινήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και μας ενδιαφέρει και η κοινωνική καινοτομία. Τέλος. Αυτό που λέτε για περισσότερη διαφάνεια. Πάντα προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη διαφάνεια, αλλά οποιοδήποτε έλεγχος από τη δικιά σας την πλευρά είναι ευπρόσδεκτος από μας γιατί έτσι μπορούμε να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη διαφάνεια. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα κύρια σχόλια που κάνατε. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μάουρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις όπως τόνισε και ε, ο πρώτος και ο τελευταίος των παρεμβενόντων πρέπει να υπάρξει ε, ε, μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης της τραπέζης να συγκεντρώνει επενδύσεις με τριπλό αλφα και από την άλλη φορά να μπορεί να επενδύσει στις περιοχές οι οποίες όντως πάσχουν στην Ευρώπη. Δεν είναι είναι ένα πάρα πολύ εύκολο πρόβλημα αλλά νομίζω ότι είναι και ο βασικός μας στόχος δηλαδή θα πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διότι θα πρέπει να μπορούμε να δεσμεύσουμε στην αγορά τα κεφάλαια τα οποία μπορούν να προωθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει βέβαια να πω ότι θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν και θα απευθυνθώ στους συναδέλφους για να τους ξαναπαρουσιάσω τις τροπολογίες με μία συνάντηση των σκιωδών εισηγητών εάν δεν μπορέσουμε να προχωρήσουμε την περίφημη τροπολογία Coffee Break του συναδέλφου Epping. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι τώρα έγινε ε, η παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως. Οι ε, τροπολογίες ε, είναι μέχρι τις 25 Οκτωβρίου για ψηφοφορία στην Επιτροπή 10 Ιανουαρίου κατά τρόπον ώστε να περάσει την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη ε, ε, ε, είναι ένα πολύ μελλοντικό, αλλά πρέπει να δούμε ποιος είναι εδώ. Είναι η έκθεση της Κέιτ, διότι αντιλαμβάνομαι ότι ο Μάρκους δεν πρόκειται να έρθει, ο Σαΐντ είναι εδώ, ο Όντι Σμιτ δεν είναι εδώ ακόμη, η Έμιλη έχει έρθει. Θα έρθει, ξέρει κανείς αν πρόκειται να έρθει. Ούτε ο Γιώργεν είναι εδώ. Οπότε και ίσως ε, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα 5-6 λεπτών μέχρι ότου να φτάσουν οι υπόλοιποι σκιώδεις εισηγητές. Λυπάμαι. Καλώς. Καταφέραμε να μαζέψουμε και μερικούς ακόμα σκιώδεις για το επόμενο θέμα μας. Οπότε ας προχωρήσουμε. Θα συστήσουμε λοιπόν τώρα τις ειδικέ απαιτήσει για τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για τροποποίηση της ε, οδηγίας. Και έχει να κάνει και με το επόμενο θέμα Φαντάζομαι η συζήτηση θα γίνει και για τα δύο μαζί. Οπότε η ΚΕΙ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντω θα συζητήσω και τα δύο θέματα, μια που είναι άρρητα συνδεδεμένα μεταξύ τους όσον αφορά την ουσία. Έχω μια αιτιολογική έκθεση που είναι νομίζω αρκετά λεπτομερής, υπάρχει μέσα στην έκθεση, οπότε θα είναι πολύ σύντομα τα σχόλιά μου, γιατί νομίζω ότι η αιτιολογική έκθεση πραγματικά σας δίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύουμε και έτσι καταλαβαίνετε γιατί έχουν γίνει τα πράγματα που έχουν γίνει. Θέλω να επιστήσω την προσοχή των Ευρωβουλευτών στο γεγονός ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι κάπως περίεργη όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Εμείς ε, ασχολιόμαστε με τις οντότητες αυτές ε, δημοσίου συμφέροντος και με την Τζούρι έχουμε επίση κοινέ αρμοδιότητε όσον αφορά τι μη ελεγκτικέ υπηρεσίε. Οπότε στην έκθεσή μου προσπαθώ να περιοριστώ στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και να μην μπω στα γενικά θέματα που έχουν να κάνουν και με τις αρμοδιότητες της τζούρι όσον αφορά τον έλεγχο. Στην ε, έκθεσή μου λοιπόν πάω λίγο πίσω σε κάτι αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη γνωμοδότηση της ΚΟΝ που ψηφίσαμε ομόφωνα ουσιαστικά για την ε, έκθεση διας πρωτοβουλίας στο φθινόπωρο που μας πέρασε. Και όσοι είχετε διαβάσει την αρχική έκθεση που είχαμε τότε και το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, θα θυμόσαστε ότι είχαμε καταλήξει στο ότι η Επιτροπή ελάχιστα πράγματα είχε συμπεριλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτά που προτείναμε εμείς και δεν συμφωνήσαμε. Τώρα λοιπόν επανέρχονται αυτά τα θέματα. Η κατάσταση στι διάφορε χώρε είναι εντελώ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Οι απαιτήσει είναι εντελώ διαφορετικέ και εφαρμόζονται και διαφορετικά. Χρειάζεται λοιπόν μια κοινή βάση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο. Στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας είχαμε επικεντρωθεί στην ποιότητα. Νομίζω λοιπόν ότι και εδώ αυτό που προσπαθώ να κάνω, ποιότητα, αυτό είναι το κύριο, το πρώτο. Τώρα πιο συγκεκριμένα στον ε, ορισμό του τι είναι οι οργανισμοί αυτοί δημοσίου συμφέροντος, οι οντότητες ε, αυτές ε, δημοσίου συμφέροντος. Εγώ πιστεύω ότι ένας έλεγχος είναι έλεγχος ανεξάρτητα με το για ποιο τύπο επιχείρησης πρόκειται. Πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική ελέγχου με ε, προϋποθέσεις που να είναι οι ίδιες, χωρίς να υπάρχει διαφορά ανάλογα με, το, με τι επιχείρηση έχουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η γραμμή μου και σε αυτήν εμένω στις τροπολογίες που προτείνω. Την ίδια λογική ακολουθώ επίσης και όταν δεν έχουμε ορισμό για τις μεγάλες οντότητες δημοσίου συμφέροντος, γιατί και πάλι λέω έλεγχος είναι έλεγχος. Η ίδια ποιότητα ελέγχου λοιπόν πρέπει να υπάρχει, είτε πρόκειται για μια μικρή οντότητα, για μια μεγάλη. Και υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Είναι να συμπεριλάβουμε πόρους στο πεδίο εφαρμογή του ελέγχου και τις απαιτήσει του ελέγχου. Θεωρώ ότι έχω κάνει πολλή δουλειά για το ERFMD και για τους ΟΣΕΚΑ. Επίσης πάρα πολλή δουλειά έχει γίνει και όσον αφορά τον έλεγχο ε, ταμείων με την νομοθεσία αυτή. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα ήταν λογικό το ERF και τους ΟΣΕΚΑ να τους δούμε σαν οργανισμούς με ειδικέ απαιτήσεις. Δεν είναι ότι εγώ πιστεύω ότι τέτοιου ταμεία πρέπει να βγαίνουν από τις απαιτήσει του πλήρους ελέγχου για να ελέγχονται οι απάτες που πολλές έχουν διερευνηθεί τελευταία. Όχι, αλλά πιστεύω ότι εμείς εδώ στην Οικονομική Επιτροπή έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά για τις καταθετικές περιπτώσεις και νομίζω ότι δεν πρέπει να με τις μεταχειριζόμαστε όπως γίνεται εδώ. Ποιος είναι ο ρόλος τώρα της ΕΣΜΑ, της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αγορών και Αξιών. Η ΕΣΜΑ έχει έναν πολύ ισχυρό ρόλο όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως ρόλο να συντονίζει και να καταλήγει σε κάποιους κανόνες και να αποφασίζει για θέματα εναρμόνισης της αγοράς που επιβάλλονται και στις 27 χώρες. Αν όμως δει κανεί προσεκτικά ποιοι κάνουν την εποπτεία του ελέγχου στις 27 χώρες μέλη, θα δείτε ότι μόνο πέντε από τις εποπτικές αρχές κινητών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την εποπτεία ελεκτικών γραφείων. Και δεν το θέλουν μάλιστα γιατί πιστεύουν ότι είναι κάτι πολύ ειδικό και ιδιαίτερο το οποίο δεν ε, διασφαλίζει τίποτα στις χώρες μέλη. Δεδομένου λοιπόν ότι η ΑΚΑ αυτή, αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή των Αξιών και Αγορών, αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, δεν θα ήταν σωστό να αποφασίσουμε για ένα ειδικό σώμα που να καλύπτει κάτι παραπάνω από τους ειδικού ελεγκτές του 25 αντί για τους 5 που έχουμε. Εξάλλου, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ομάδα Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών που υπάρχει ήδη για την διαχείριση αυτών των καθηκόντων που θέλει να αναθέσει στην ΕΑΚΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι βέβαια επίπεδου 3 επιτροπή, οπότε δεν μπορεί να έχει ακριβώς τις ίδιες ε, αρμοδιότητες όπως έχει η ΑΚΑ. Γι' αυτό με τις τροπολογίες μου προσπαθώ να τους δώσω όσο γίνεται περισσότερες αρμοδιότητες, ενώ στο νομικό πλαίσιο θα έπρεπε να έχουν συμβουλευτικό ρολόγο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το πάω και λίγο ακόμα πιο μακριά. Πιστεύω ότι ο ΕΟΦΕ θα μπορούσε να είναι Επιτροπή Λομφαλουσί. Και νομίζω ότι έτσι το καταλαβαίναμε για χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να έχει περισσότερες εξουσίες. Αλλά εξαρτάται και από το Συμβούλιο, γιατί το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο θα αποφασίσει αν θέλει Επιτροπή Λομφαλουσί για τον έλεγχο ή όχι. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια των συναδέρφων εδώ να μου πούν αν θέλουν να προχωρήσουμε έτσι ή όχι. Οπότε το θέμα δεν είναι αν θέλουμε συντονισμό ή έλεγχο από ένα ευρωπαϊκό σώμα, είναι να βρούμε ποιο είναι το κατάλληλο ευρωπαϊκό σώμα που έχει την δυνατότητα και την πραγματογνωμοσύνη για να εφαρμόσει μια αναρμονισμένη διαδικασία ελέγχου και στις 27 χώρες. Τώρα έρχομαι στον διάλογο με τους εθνικούς ελεκτές. Σύμφωνα με την οδηγία για τι κεφαλαικέ απαιτήσει την 2, ο διάλογο αυτό με του εθνικού ελεγκτέ θα έπρεπε ήδη να λαμβάνει χώρα. Όμω, σε πολλές χώρες μέλη δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Οι ελεκτές δεν είναι βέβαια επόπτες, μπορούν όμως να συμβουλέψουν για τις πρακτικές στην αγορά. Και νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα κάτι που παραδέχονται όλοι, ότι μπορεί να υπάρχει μια διπλής κατεύθυνση σχέση ανάμεσα στους ελεκτές και τους επόπτες, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται σε ορισμένα δημοσιονομικά ιδρύματα και τομείς που είναι κλειδί. Θα έπρεπε επίσης να κάνουμε και ένα άλλο βήμα, να έχουμε και μια ε, τριπλής κατεύθυνσης διαδικασία, να υπάρχει δηλαδή συμμετοχή και στο διάλογο πολλές φορές προτείναμε ότι αυτά πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση. Να υπάρχει ένα τέτοιο φόρουμ, τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο. Άρα να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου να καθορίζεται πότε θα λαμβάνει η χώρα αυτός ο διάλογος. Έτσι θα έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις μέσα στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Διάλογο λοιπόν λέμε με τους εθνικούς ελεγκτές τότε πρέπει ο διάλογος να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τομέα. Τώρα έχουμε μεν την ACIB, αλλά είναι βασική σημασία όσοι γνωρίζουν τους τομείς, ιδιαίτερα στις δημοσιονομικές υπηρεσίες, να μπορούν να βοηθούν για να καταλαβαίνουμε καλύτερα ποιες είναι οι τάσεις ανώνυμα βέβαια. Πάντως ο ρόλος των ελεγκτών είναι να είναι επαγγελματίε που να εκτιμούν κατά πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει περίπτωση για συστημικό κίνδυνο. Ένα τέταρτο θέμα που θέλω να αναπτύξω εδώ είναι ο ανταγωνισμός. Στην ε, πρώτη έκθεση πρωτοβουλίας συζητούσαμε πολύ για τον ανταγωνισμό και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον ε, ανταγωνισμό σε σχέση με τον έλεγχο. Για τις περισσότερες από τις μεγάλες επιχειρήσεις η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πάνω από τέσσερις επιχειρήσεις που αναμειγνύονται για τον έλεγχο. Χρειάζονται όμως μέτρα τα οποία να εξετάσουν τη δομή της αγοράς και να βασίζονται σε μια ανάλυση ωφέλους και όχι απλώς να επιβαρύνουμε παραπάνω κόστος στις επιχειρήσεις που θα ελεγχθούν δεν γίνεται να υπάρχει ένα τέτοιο δυσανάλογο κόστο σήμερα στην περίοδο κρίση που περνάμε, γιατί δεν υπάρχει όφελο τελικά ούτε για τι επιχειρήσει ούτε για την κοινωνία ολόκληρη. Δεδομένου λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει νέα στοιχεία για μια μελέτη κόστου ανάλυση και δεν υπάρχει τίποτα που να μα επιβεβαιώνει για το όφελο, εκφράζω την ανησυχία μου. Ένας υποχρεωτικός και τακτικός έλεγχος μήπως είναι περί το κόστος. Και όσοι από εσά γνωρίζετε καλά τις οικονομικές αυτές επιχειρήσεις, πολλές από αυτές έτσι κι αλλιώς έχουν που πρέπει να αντιμετωπίσουν, το οποίο από μόνο του σημαίνει ότι επιβαρύνονται με ένα επιπλέον μεγάλο κόστος. Συνεπώς, να διατηρήσουμε την ποιότητα του ελέγχου αλλά να μην αυξάνουμε το κόστος για να αυξήσουμε το κόστος και μόνο. Εγώ έχω καταλήξει και σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα όσον αφορά τους διαγωνισμούς και την υποβολή προσφορών. Μια υποχρεωτική υποβολή προσφορών θα ήταν κάτι θετικό γιατί τότε σε τακτική βάση ε, οι υπηρεσίες ε, αυτές θέτουν το ερώτημα κατά πόσο έχουν τις καλύτερους ελέγχους, κάτω από τους καλύτερους όρους. Εγώ προσωρινά ο κοινό έλεγχο δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά. Από την άλλη όμω το να ενθαρρύνουμε τον επιμερισμένο έλεγχο είναι κάτι που αξίζει τον κόπο. Και πιστεύω ότι ενώ μια επιχείρηση παίρνει την ευθύνη για μια ολόκληρη ομάδα, άλλες επιχειρήσεις ελέγχου ελέγχουν τις θηγατρικέ του και μερικέ φορέ θηγατρικέ κλειδί από διαφορετικέ επιχειρήσει. Με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούν τον ελεγκτικό τους ρόλο. Αλλά αυτή είναι μια απόφαση που γίνεται ανά επιχείρηση και καταλήγουν ε, μετά σε συμπέρασμα για το αν είναι αυτό καλό ή όχι. Εγώ δεν θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει υποχρέωση να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και ένα άλλο κερδοσκοπικό στοιχείο για τις ελεγκτικές επιχειρήσεις είναι οι μη ελεγκτικές ε, επιχειρήσεις. Υπάρχουν απογορεύσεις σε αυτό, αλλά υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που επιτρέπεται να δρουν μέσα σε αυτό το σύστημα. Την υποβολή προσφορών πρέπει να την ξαναδούμε. Πόσο κερδοσκοπικό είναι αυτό. Μήπως θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε τις μικρές ελεκτικές επιχειρήσεις να συνεργάζονται με τις μεγάλες και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Έτσι θα βοηθηθούν όταν υποβάλλουν προσφορές για μεγαλύτερους ελέγχους να, είναι, να έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν το στόχο τους. Ο τελικός σκοπός στη διαδικασία υποβολής προσφορών είναι να δώσουμε μεγαλύτερη δύναμη στις ελεγκτικές επιτροπές. Αυτές πρέπει να εξετάζουν τη δουλειά που γίνεται όσον αφορά τους ελέγχους και να αξιολογούν την ποιότητα προς όφελος ολόκληρης της επιχείρησης που ελέγχουν και ολόκληρης της κοινωνίας. Μια ισχυρή ελεγκτική επιτροπή με καλό έλεγχο και αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου είναι θεμελιώδης σημασίας. Αυτά προσπαθώ λοιπόν να υπογραμμίσω στην έκθεση αυτή. Τώρα αν υπάρχουν ε, σχόλια ευχαρίστω να τα ακούσω γιατί αυτή είναι μια διαδικασία χωρίς τέλος, με την οποία προσπαθούμε να πετύχουμε όσο γίνεται ευρύτερη συνένεση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο Μάρκος μου είπαν ότι δεν θα μπορέσει να έρθει. Και δεν νομίζω ότι έχει ζητήσει από κάποιον να τον αντικαταστήσει, εκτός αν υπάρχει κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο αυτού. Αλλιώς ο Σαΐντ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια είναι μια καλή βάση προς συζήτηση η έκθεση αυτή. Σίγουρα δεν συμφωνούμε με όλα. Θυμάμαι την αρχική πρόταση. Συμφωνούμε για το ότι η κρίση κατέδειξε ότι η ποιότητα του ελέγχου πρέπει να βελτιωθεί. Με διάφορους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Υπάρχουν οι προτάσεις κείμενο που έχουμε στη διάθεσή μας. Για μας πάντως ο στόχος πρέπει να είναι πώς μπορούμε όσο γίνεται με περισσότερη ακρίβεια να πετύχουμε τον σωστό έλεγχο μιας επιχείρησης έτσι ώστε οι επενδυτές να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη. Άρα ο ρόλος των ελεκτών είναι τεράστια σημασίας. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα εδώ είναι η αρχή του εκπεριτροπής ελέγχου. Έχω την εντύπωση ότι αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για να αλλάξει η δομή, αλλά αν θέλουμε τέτοιον εκπεριτροπής έλεγχο, τότε δεν θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος αυτός να περιορίζεται μέσα σε ένα κύκλο ελεγκτικών ε, εταιριών. Θα πρέπει να διευρύνεται. Άρα αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Κάθε πόσα χρόνια θα γίνεται η αλλαγή, για παράδειγμα. Αυτό που προτείνεται, μήπως είναι λίγο. Επίσης, ένας συνδυασμός με το σύστημα των μεικτών ελέγχων. Joint audits. Θα έπρεπε σαν προϋπόθεση να έχει ότι κάθε τόσο γίνονται πολύ σοβαροί έλεγχοι. Και σε τι ποσοστό, 40, 60, 50, 50. Διάβασα βέβαια αυτά που λέτε για τις εναλλακτικές στους μεικτούς ελέγχους. Πάντως η αρχή να είναι διαφορετικές οι επιχειρήσεις είναι μια υγιής αρχή και μειώνει το περιθώριο λάθους ή κινδύνου. Τώρα τι υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει η ελεγκτική εταιρεία. Υπάρχει ο κίνδυνος, αν ε, είναι πολλές ε, ιδέες που συμπεριλάβουμε εδώ, να μειωθεί η ποιότητα. Η εισηγήτρια κάνει πάντως διάφορες προτάσεις. Κάθε σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να αποκλειστεί πάντως, όπου και αν καταλήξουμε και να έχουμε εγγυήσει. Συνεπώς, η πρόταση της εισηγήτριας πιστεύουμε ότι είναι επαρκής, παρόλο που θα κάνουμε και κάποιες προτάσεις για να ενισχυθεί η πρότασή της. Το θέμα τώρα της εποπτείας του ελέγχου. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό διαρθωτικό στοιχείο που πρέπει να βελτιωθεί. Άρα χρειάζεται ο διάλογος με τους εθνικούς ελεκτές Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία. Εδώ τίθονται σοβαρά ερωτήματα και υπάρχει από τον κλάδο μεγάλος σκεπτικισμός όσον αφορά την ανεξαρτησία τους. Σίγουρα χρειαζόμαστε μια ισχυρή εποπτεία στην Ευρώπη και είμαστε έτοιμοι μαζί με την εισηγήτρια να το συζητήσουμε αυτό και να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις. Πάντως είπαμε ότι η βάση είναι να έχουμε και να οργανώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλό έλεγχο με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τους εθνικούς ελεκτές. Για την Ελεγκτική Επιτροπή, αυτά που λέτε είναι ένα βήμα προς τα μπρος, συμφωνούμε μαζί σας, η Επιτροπή αυτή, η Ελεγκτική, θα πρέπει όντως να έχει ανεξαρτησία από το Διοικητικό Συμβούλιο, να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και να κρίνει την ποιότητα των ε, εποπτικών εκθέσεων. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τον έλεγχο και την εποπτεία γενικώ για τα στοιχεία των ε, εταιριών που έχουμε στη διάθεσή μας. Χρειάζονται αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, οπότε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια καλή βάση. Έχει προσθέσει μερικά θετικά και η συγγήτρια και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά πιστεύουμε ότι θα συνεργαστούμε επικοδομητικά με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Ε, ρωτώ τους ε, σκιώδεις. Ε, Ζων Πολ νομίζω ότι ζήτησες να μιλήσεις τελευταίος και έτσι τώρα είναι όλοι Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κέι. Εξαιρετική έκθεση ως συνήθως. Ε, βεβαίως ε, παρόλο που το, Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην ε, νομισματική ένωση έχει, έχει σταυμάσιες ιδέες. Βέβαια είναι μια πολύ ουσιαστική έκθεση και θα πρέπει να την εξετάσουμε από την οπτική γωνία των χρηματαγορών και των ρυθμιστικών ε, μεταρρυθμίσεων και των προβλημάτων. Οπότε όλοι συμφωνούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει από αυτού. Αλλά το θέμα είναι ε, πώς και ποιος είναι ο τρόπος. και είπες ότι το βασικό είναι η ποιότητα του ελέγχου και πόσο θα μπορέσει να επεκταθεί ε, η εντολή ε, των οικονομικών ελεγκτών. και ε, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα των σχετικών εκθέσεων διότι πιστεύω ότι όλοι έχουμε πιεστεί και προσεγγιθεί τις τελευταίες, τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, αλλά είμαστε λογικοί. Ξέρουμε ότι η ποιότης πρέπει να βελτιωθεί. Το, το τι, πώς θα επιτευχθεί αυτό είναι αμφισβητήσιμο. Ε, <clears throat> όσον αφορά τον κανονισμό. Εγώ έρχομαι από μια μικρή χώρα, ξέρω ότι η Σιλβή δεν θέλει να το αναφέρω, αλλά έτσι είναι. Επειδή λοιπόν η χώρα μου είναι μικρή, εάν υπάρξει ένας κανονισμός μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μία οδηγία η οποία θα βασίζεται στις αρχές. Ξέρω ότι δίστανται οι γνώμες, αλλά έχουμε διαφορετικές μεθόδους επιλύσεως αυτών των θεμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν απόψεις που συγκρίνονται με τις ε, προτάσεις. Ε, παραδείγματος χάρη με τον τρόπο που εμείς το ε, συζητάμε στη χώρα μας και πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, ε, παραδόσεις ως επιχειρήσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτές οι διαφορές θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Δεν πιστεύω ότι όλοι μπορούν να μπουν σε ένα καλαπόδι και αυτό θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται και στην πρόταση. Έχω να κάνω και άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την ε, κοινή, ε, τον κοινό οικονομικό έλεγχο. Πιστεύω ότι ε, θα αυξήσουμε και το κόστος και το βάρος. Εάν πρέπει να υπάρχει μία εναλλαγή στον, μία ναι, μια εναλλαγή στον έλεγχο, αμφισβητήσιμο, ε, ανταγωνισμός της αγοράς. Όντως χρειάζεται και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων εταιριών. Ε, δεν ξέρω όμως πώς θα το επιτύχουμε. δεν ξέρω αν αλλάζοντας ε, τον κανονισμό ή την οδηγία μπορούμε να το επιτύχουμε ή αν αυτή είναι η μόνη λύση. Οι εταιρείε αυτές θα πρέπει βέβαια να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν αλλά θα πρέπει να αξιολογούνται με πολύ προσεκτικά κριτήρια. Πιστεύω ότι η βασική αρχή είναι ότι θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να αποφασίζουν πότε πρέπει να αλλάξουν ελεγκτές ε, και πότε θα πρέπει να αλλάξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν συγκρόμενα συμφέροντα και είμαι σκεπτικός σχετικά με την εναλλαγή, τη rotation που προτείνεις. Ε, Σα δεν σε κατάλαβα. Δεν, δεν κατάλαβα δηλαδή αν εσύ ήσουν υπέρ ή κατά αυτής της μεθόδου. Θα το συζητήσουμε, εντάξει. Αμφισβητώ επίσης και την υποχρεωτική, τον υποχρεωτικό διαγωνισμό διότι δημιουργείται κόστος και για τις εταιρείες και για τις ελεγκτικές εταιρείες ε, διότι υποχρεωτική, ο υποχρεωτικός μειοδοτικός διαγωνισμός κάθε έξι χρόνια έχει και μειονεκτήματα. Ένα τρόπος ήταν να υποχρεώσουμε τις εταιρείε ε, ελεγκτών να ε, δημιουργήσουν ε, ένα μηχανισμό εναλλαγής τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια με πλήρη διαφάνεια προς τους μετόχους. Επίσης όσον αφορά την πιστοποίηση που είναι ένα θέμα το οποίο διέγραψες και θα σε παρακαλούσα να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο. Διότι πιστεύω ότι η ιδέα αυτή είναι καλή. Όσον αφορά το ε, άρθρο σχετικά με την ύπαρξη ή όχι του οικονομικού ελέγχου, ε, θα χρειαζόταν η ε, ρητή άδεια της Επιτροπής Ελεγκτών. Κατά τη γνώμη μου, Εάν ζητάμε ε, να γίνει ένας έλεγχος εάν καλύπτεται το 10% της ε, αμοιβή των ελεγκτών είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω. Εάν μπορούν να αναλάβουν και ε, άλλα καθήκοντα θα πρέπει να προσέξουμε να διατηρηθεί η διαφάνεια και γι' αυτό και πρέπει να ελέγχουμε ποιες θα είναι οι αμοιβέ για τους οικονομικούς ε, να υπάρχει μεγαλύτερη ε, ανταγωνισμός όσον αφορά τη διαφάνεια και τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Και τέλος η εποπτεία. Ε, είμαστε υπέρ του ΕΣΜΑ αλλά δεν μπορώ να ακολουθήσω το σκεπτικό της και εδώ και ίσως θα έπρεπε ΕΟΦΕ, το ΕΟΘΕ να μεταμορφωθεί σε ένα πρότυπο το οποίο ε, θα είναι υπόλογο. Αυτό θα ήταν μία λύση και σας ευχαριστώ. Thank you. Ε, Emily. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για τις δύο αυτές εκθέσεις. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι οι πράσινοι συνεργαστήκαμε με τους συναδέλφους σας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μπορώ να σχολιάσω το σύνολο λοιπόν της προσπάθειας, αν και υποτίθεται εδώ στην οικονομική είμαστε κάπως πιο περιορισμένοι σε σχέση με τους στόχους που έχουμε, αλλά οι, αντικα... οι τροπολογίες των συναδέλφων αντικατοπτρίζουν, θα έλεγα, το σύνολο της προβληματικής και στις δύο εκθέσεις. Όπως είπε και ο Σαΐντ, η χρηματοοικονομική κρίση δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στον τομέα του λογιστικού ελέγχου. Υπάρχουν προβλήματα ποιότητα, συγκρούσεων συμφερόντων και βλέπουμε και πάρα πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις στην αγορά. Αυτά τα τρία θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν δούμε την έκθεση Swinburne και την έκθεση της Jury, δεν νομίζω ότι είναι επαρκείς οι προτάσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία παραμένουν. Η έκθεση της Επιτροπής ήταν γενναία εν πολλής. Μπορούμε να συζητήσουμε κάποιες από τις λεπτομέρειές της, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για να μην φανούμε υπερβολικά επιφυλακτικοί. Απαιτείται λοιπόν ε, στα τρία θέματα που προανέφερα να είμαστε κάπως ε, πιο ε, θαραλέοι και να μην μείνουμε, να μην αρκεστούμε στο status quo. Απαιτείται μια δυναμική και ανταγωνιστική αγορά με περισσότερους παίκτες. Απαιτείται καλύτερος έλεγχος και εποπτεία με στόχο τη βελτίωση του λογιστικού ελέγχου και την έβρεση των μέσων τα οποία είναι ανάλογα και επαρκή για να βελτιωθεί η κατάσταση. Η εναλλαγή είναι μία δυνατότητα, δεν το αποκλίνουμε. Θα δούμε κάθε πόσα χρόνια, αλλά είναι σίγουρα ένα μέσο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Έχουν γίνει και άλλες συζητήσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Είναι δύσκολο να περάσουμε σε πλήρη εναλλαγή, ε, αλλά είναι μία δυνατότητα. Υπάρχει επίσης ε, δυνατότητα για κίνητρα έτσι ώστε να υπάρχουν από κοινού ε, λογιστική έλεγχη. Ε, κίνητρα στον τομέα των προμηθειών, των διαγωνισμών μάλλον δεν είναι επαρκή από μόνα τους. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις της Επιτροπής, αλλά το θέμα των διαγωνισμών δεν θα λύσει από μόνο του το θέμα της έλλειψης επαρκούς αριθμού παικτών σε εισαγωγικά στο λογιστικό έλεγχο. Θα πρέπει να επιτρέψουμε επίσης και σε μικρότερες εταιρείες ορκωτών λογιστών να μπουν στην αγορά και να σπάσουμε την ολιγοπολιακή κατάσταση η οποία σοβεί σήμερα. Θα πρέπει παράλληλα να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αύξησης λοιπόν των ε, παικτών με θετικό τρόπο. Ένα τελευταίο σημείο για σήμερα τουλάχιστον. Σαν σημείο εκκίνησης εμείς θα εξετάσουμε σε βάθος ε, την πρότασή σας. Είμαστε εμείς υπέρ της ΕΣΜΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν επιπλέον πόροι βέβαια. Πρόκειται για ένα σώμα το οποίο ήδη έχει πάρα πολλά να κάνει και το πρόβλημα είναι ότι ε, μονίμως θα έλεγα ε, χαρακτηρίζεται από έλλειψη πόρων. Αλλά αν δώσουμε περισσότερες δυνατότητες ελέγχων στην ΕΣΜΑ θα πρέπει να ενισχύσουμε και τους πόρους που έχει στη διάθεσή της. Έχετε όμως και διαφορετικά επιχειρήματα για το ποιο θα είναι το καλύτερο μέσο και σώμα για αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Εμείς έχουμε άλλες απόψεις. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα κοινό και ισχυρό ευρωπαϊκό σώμα που να ελέγχει το κλάδο του λογιστικού ελέγχου. Δεν θα περάσω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία με τους κοιόδης. Ελπίζω να γίνει αυτό το γενναίο βήμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την κρίση. Ευχαριστώ. Ο Κλούτε δεν είναι εδώ, οπότε έχει το λόγο ο Γκοζές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ακουστώ διαφορετικά από ό,τι ακούστηκε μέχρι τώρα τουλάχιστον μας λέγουν ότι ο λογιστικός έλεγχος είναι αυτός που είναι και οι ελλείψεις λογιστικού ελέγχου είναι μία από τις αιτίες της κρίσης που βιώνουμε. Παραδείγματα δώστε μου. Στον τομέα του λογιστικού ελέγχου υπάρχουν τρομερές διαφορές από τη μια χώρα στην άλλη. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις ακόμα και στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πρακτικής ε, ε, είναι διαφορετικές και υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λογιστικού ελέγχου. Στόχος του λογιστικού ελέγχου, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι να προλαμβάνει κρίσεις, αλλά να ελέγχει την ομιμότητα των λογαριασμών, την αυθεντικότητά τους και τον ένομο χαρακτήρα τους. Ήδη λοιπόν θα πρέπει να φανούμε εδώ να δείξουμε κάποιο μέτρο αν και γενικότερα δέχομαι τις προτάσεις του Επιτρόπου, θα πρέπει να φανούμε πραγματιστές. Πολλοί από αυτούς που μιλούν για τα θέματα του λογιστικού ελέγχου δεν έχουν δει πώς δουλεύουν οι ορκωτοί λογιστές, δεν είχαν επαφές μαζί τους και η κατάσταση όπως σας είπα δεν είναι αυτή η καταστροφή την οποία περιγράφουν οι περισσότεροι. Υπάρχουν ορισμένε λοιπόν προτάσεις τη επιτροπή για τη βελτίωση του λογιστικού ελέγχου. Τόσο το καλύτερο, γιατί όχι εφόσον το μπορούμε, αλλά και εδώ να θέσουμε το θέμα ε, ποιο είναι το σημείο εκκίνησης. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, δεν ήμασταν σε ζούγκλα, υπήρχε μία κάποια ποιότητα. Και σε κάποιες προτάσεις που γίνονται πρέπει να σταθούμε λίγο <clears throat> για τις κοινέ δραστηριότητες ελέγχου. Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα με, αυτό το, με χώρες όπου υπάρχει το λεγόμενο συνδυασμένο σύστημα ορκωτών ελέγχων. Δεν είναι δύο εταιρείε, αλλά είναι από τέσσερις τομείς που ασκείται ο έλεγχος και δεν μιλάμε για μια κατανομή που θα μπορούσε να λειτουργήσει σε όλες τις χώρες. Μας λέτε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το επιπλέον διοικητικό κόστος και γραφειοκρατικό κόστος. Θα πρέπει να δούμε εδώ τη σχέση κόστους και ωφέλους και θα πρέπει να δούμε ότι εκεί που αυτή η πρακτική, όχι ο συνδυασμένος ε, ορκωτός έλεγχος, αλλά ο ε, συνδυασμένος ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα ελέγχου. Σε κάποιες χώρες ε, είναι απαραίτητο αυτό το σύστημα για τις επιχειρήσεις στη Γαλλία σαν παράδειγμα που είναι στις 40 μεγαλύτερες του χρηματιστήριου και στις τράπεζες. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει, ε, θα έλεγα, ε, ανταγωνισμός. Έχουμε τέσσερις μεγάλες εταιρείες ορκωτού ελέγχου που θέλουν να σκοτώσουν όλους τους υπόλοιπους. Και αν οργανώσουμε την εναλλαγή θα εναλλάσσονται μεταξύ τους. Δεν θα επιτρέψουν στους μικρούς τους οποίους θα τους συντρίψουν. Και εδώ τίθεται σε αμφισβήτηση η αρχή της εναλλαγής που καταπολέμησα ε, εγώ στο σύστημα των ε, εταιριών αξιολόγησης γιατί αντί για τρεις μεγάλες που έχουμε σήμερα θα μας είχαν εξεμείνει δύο. Λοιπόν, και θα πρέπει να δούμε επίσης και το κόστος όπως της εναλλαγής, όπως είπε ο Σμίτ για τις επιχειρήσεις. Εγώ τα έχω κάνει αυτά και αν πρέπει κάθε 5-6 χρόνια να ψάχνουμε για καινούριε εταιρείε ορκωτών λογιστών, αυτό θέλει χρόνο, κοστίζει και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι οι νέε εταιρείε ορκωτών λογιστών θα είναι αποτελεσματικότερε των προηγούμενων. Βέβαια, θα πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα κλειστά συστήματα. Στην Γαλλία, α πούμε, έχουμε αυτό το σύστημα με τα τρία χρόνια. Και εδώ χρειάζεται ένας μέσος όρος για τις επιτροπές ελέγχου θα πρέπει εδώ να φανούμε προσωπικοί. Ε, δεν μιλάμε για υπερελεγκτές εδώ, πρόκειται όμως για ένα ειδικό επίπεδο ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολείται με τον λογιστικό έλεγχο αλλά θα πρέπει να λέμε ότι, εξ αυτού ότι ο έλεγχος θα πρέπει να ασκείται προς τους ορκωτούς λογιστές. Αυτό σημαίνει ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι ε, ένα μεγάλο κομμάτι του ορκωτή λογιστές. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Γιατί τότε θα πρέπει σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο μιας μεγάλης επιχείρησης να υπάρχουν ειδικοί τους, ε, για τον λογιστικό έλεγχο, ε, για τα οικονομικά, για τα οικονομετρικά, για τα πιστοτικά κτλ. Οπότε αλλάζουμε εντελώ οικονομική δραστηριότητα. Τώρα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου και μη λογιστικού ελέγχου. Εδώ μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις συμφερόντων. Αν δούμε προσεκτικά τα πράγματα θα δούμε ότι στα πλαίσια των δευτερευουσών υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται υπάρχει θα έλεγα μια διασταυρούμενη γονιμοποίηση. Τι εννοώ με αυτό. Θα πρέπει οι ελεγκτές να προσπαθήσουν να βρουν το πρόβλημα της επιχείρησης. Για να το πετύχουν πρέπει να είναι στην πραγματικότητα. Αλλιώς θα είναι ψυχροί παρατηρητές που δεν αναγνωρίζουν παρά μόνο αυτά τα οποία τους δίνουν και που μερικές φορές ε, δεν βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, τα κόλπα που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να παρακάμψει κάποιες ρυθμίσεις ή για να μακιγιάρει κατά κάποιο τρόπο τους λογαριασμούς της επιχείρησης. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε μια σωστή διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο είδη δραστηριοτήτων έτσι ώστε οι δευτερεύουσες αυτές οι υπηρεσίες να μην παρέχονται από τις υπηρεσίες που, που ασκούν αυστηρά τον λογιστικό έλεγχο. Ο Μάρκους Φέρμπερ εδώ θα συνέχερε την εισηγήτρια για την εργασία της και αυτό ακριβώς κάνω και εγώ. Σάιμον, Σίμον μάλλον. Από δική μου πλευράς θερμές ευχαριστίες για αυτή την πρόταση που είναι μια καλή βάση συζητήσεως και ιδίω η πρόσκληση για υποβολή μειοδοτικών προτάσεων. Ήθελα όμως να αναφερθώ σε διάφορα σχόλια. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, με ενδιέφερε πάρα πολύ να συζητήσω με επιχειρήσεις της δικιάς μου περιφέρειας όπου είναι οι μεγαλύτερες ε, οι ε, εταιρείε της Γερμανίας και ασχολόμουν με το θέμα πριν εκλεγώ το 2009 και βλέπω ότι οι μεγαλύτερες ε, εταιρείε είναι επιφυλακτικές γιατί όσο αυξάνονται αυτοί οι οικονομικοί έλεγχοι αντιλαμβάνεται κανείς πόσο περίπλοκοι γίνονται. Επίσης, εάν είναι πολύ μεγάλη η επιχείρηση κάποιος θέλει να ελέγχεται από έναν. Δηλαδή ε, πρέπει να έχει από, μία, από έναν ελεγκτή και, τις, ε, και τα υποκαταστήματα και ε, όλες τις θηγατρικές εταιρείες. Όταν αντιληφθεί κανείς το περίπλοκο αυτό χαρακτήρα του ελέγχου και το συγκρίνει με τα προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει σε εταιρείε οι οποίες είχαν επί για τον ίδιο ελεγκτή και άλλαξαν προσφάτως και δούμε πόσος χρόνος χρειάστηκε από πλευρά της επιχειρήσεως για να υπάρξει η ίδια ποιότητα ελέγχου με αυτόν που είχαν στο παρελθόν λόγω του που χαρακτήρα και της ε, διασποράς σε ολόκληρη την υφίλιο, τότε χρειάζονται προθεσμίες οι οποίες θα πρέπει να είναι μάλλον ε, μεγαλύτερες από ό,τι μικρότερες. Από ό,τι κατάλαβα δηλαδή έξι χρόνια για τέτοιες μεγάλες εταιρείες μπορεί κανείς ε, να θεωρήσει ότι μπορεί να υπάρξει ε, να επιτύχει κανείς ένα σωστό έλεγχο οπότε τότε θα αναρωτηθούμε εάν επιτέλους μπορεί μια επιχείρηση να ελεγχθεί ικανοποιητικά και εξαιρετικά γιατί να αλλάξουν ακριβώς εκείνη τη στιγμή οπότε χάνουμε την απόδοση των εργασιών που έχουν γίνει κατά 6-7 χρόνια. Θα έπρεπε λοιπόν να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και να μην ξεχνάμε αυτή την οπτική γωνία. Επιπλέον χρειαζόμαστε και εδώ ευχαριστώ την εισηγήτρια την εναλλακτική λήξη να υπάρχει μια αλλαγή ε, όχι με μια ανακύκλωση αλλά να ελέγχονται κάποια στιγμή ένας αριθμός μειοδοτικών προσφορών κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσουμε να υποχρεώσουμε την Επιτροπή Ελεγκτών να ε, ελέγξουν τι άλλες ε, προσφορές υπάρχουν και αν κάποιος παραμείνει με τον ίδιο οικονομικό ελεγκτή να δει για γιατί το πράττει και δεν αλλάζει. Δηλαδή υπάρχουν τεχνικές εναλλαγές τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό που είναι βασικό για μένα είναι καταρχήν το θέμα της, όχι τόσο πολύ της εναλλαγής ε, αλλά να δούμε ε, ποιο είναι το μέγεθος των εταιριών τις οποίες θέλουμε να ελέγξουμε και νομίζω το μέγεθος αυτός ξεφεύγει από αυτό που είχε λάβει υπόψη στην Επιτροπή όταν κατήρτισε την πρόταση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να παρέμβει και έτσι έχω ορισμένε παρατηρήσεις. Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω πολλά τα θέματα που πραγματεύεται η έκθεση. Σε ορισμένα θέματα υπάρχουν, ε, ε, έχω διαφορετικές απόψεις ή χρειές σχετικά με τις υπηρεσίες που δεν είναι οικονομική έλεγχη. Είχαμε το ε, θέμα αυτό τον Ιούλιο στη Μεγάλη Βρετανία ο όπου ε, ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο είπαν ότι θαυμάζουν τους Ευρωπαίους ε, ελεγκτές και δεν θα ήθελαν να περιοριστούν μόνο στον οικονομικό έλεγχο διότι οι πιο έξυπνοι θέλουν να προσφέρουν και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες. Με συγχωρείτε αλλά φτανίζομαι λέει η πρόεδρος και συμφωνούν με τον κίνδυνο να υπάρξει μία καταστολή ε, αν περιορίσει κανείς τις ελεκτικές εταιρείες. Ίσως κάποιος τους έσπρωξε ίσως να πούν κάτι τέτοιο αλλά αυτοί αντελήφθηκαν ότι ήταν η πείρα τους και συμφωνώ ότι πολλές ε, ε, δραστηριότητες μη ελεγκτικού χαρακτήρα θα πρέπει να διατηρηθούν και να γίνονται άλλων ειδών έλεγχοι σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι όχι. Αυτό που με ενδιαφέρει σχετικά με τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες οικονομικών ελεγκτών είναι ότι ελέγχουν, συμβουλεύουν και ε, προτείνουν και πιέζουν. Νομίζω λοιπόν ότι πολλές φορές ε, το παρακάνουν. Δηλαδή αν ε, τα κάνουν όλα ε, είναι κάπως δυσαρεστό και θα έπρεπε να το λάβουμε υπόψη μας. Σχετικά με το ρόλο της ΕΣΜΑ. Ε, αντιλαμβάνουμε το πρόβλημα και προσπάθησα να το λύσω σχετικά με το, τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου διότι ορισμένες επιτροπές του μηχανισμού αυτού ε, ε, μπορούν να οδηγήσουν στο να ακολουθεί ο ελεγκτής και μπορώ να δεχθώ την πρότασή σας αν είναι κάποιος ο οποίος απουσιάζει επί μακρύ χρονικό διάστημα αλλά υπάρχει κάποια ε, διάταξη σχετικά με αυτό και για τις τράπεζες ή τους μεγάλους οργανισμούς που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως αφού μας ενδιαφέρουν οι τράπεζες μιλάμε για ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα και μιλήσατε και για το ESRB και την ε, ανάλυση οποία θα γίνει μέσω της ίσης και πάλι θα πρέπει να υπάρχει διάλογος μεταξύ των ε, υπευθύνων και θα πρέπει ε, πάντοτε ε, αν όχι να μπορούν να μιλάνε οι ελεκτές με τους νομοθέτες και όχι υποχρεωτικά και οι τρεις μαζί και όχι μόνο αυτούς που ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά και χρηματιστικά θέματα και ε, να μιλάνε με την ESRB. Οπότε ε, το, το ΕΣΜΑ έχει ένα ρόλο εδώ, αλλά εσείς είπατε ότι έχει ρόλο και το EGAOB ε, το οποίο είναι πιο κρίσιμο ίσως σε ορισμένους από ό,τι στους άλλους. Και σχετικά με το θέμα αυτό πιστεύω ότι εάν δεν αναφερθεί η πτυχή αυτή στο αίσθημα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Εγώ ήμουν θετική για την, τον κοινό έλεγχο και ε, θα υπήρχε μια λύση συνδυασμένων ενασγάτων και ποινών. Δηλαδή ε, θα, να υπήρχε ενθάρρυνση για ε, κοινό έλεγχο αλλά τελικά ε, καλύτερα να υπάρχει εναλλαγή ίσως θα πρέπει να διευρύνουμε την περίοδο σε 14 χρόνια γιατί εάν κανείς οργανώνει μειοδοτικό διαγωνισμό είναι καλό και εγώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχω ορίσει ελεγκτές και στην Αγγλία και εδώ με μια διαδικασία ε, ε, εθελοντικών προσφορών και όχι υποχρεωτικού μειοδοτικού διαγωνισμού όλοι ε, ήταν ε, ε, όλες οι προτάσεις ε, ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα και εγώ ετάραξα τα ύδατα διότι δεν πήρα αυτόν τον οποίο είχαν συμφωνήσει να προωθήσουν αλλά θα πρέπει και εμείς να ελέγξουμε και να δούμε τι θέλουμε να επιτύχουμε με τον οικονομικό έλεγχο. Έχουμε νέες ιδέες σχετικά με ορισμένα πράγματα τα οποία πιστεύουμε μπορούν να γίνουν με τον ένα τρόπο και βλέπουμε να γίνεται με ένα διαφορετικό. Άρα οι επιτροπές οικονομικού ελέγχου θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτή τη διαδικασία ε, των μειοδοτικών διαγωνισμών κατά διαστήματα όχι συνέχεια γιατί είναι μια δαπανηρή διαδικασία, αλλά μιλάμε για μεγάλες ε, μονάδες δημοσίου συμφέροντος, οπότε όταν πρόκειται για μεγάλες εταιρείε δημοσίου συμφέροντος νομίζω ότι ε, αντέχει η τσέπη τους και αν ε, ζητούσαμε μία εναλλαγή κάθε 14 χρόνια υπάρχει αρκετός καιρός να προετοιμαστούν και εντωμεταξύ να γίνεται ένας έλεγχος ή, ή στο μέσον υποχρεωτικός μειοδοτικός διαγωνισμός κατά τρόπον ώστε η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου και η δικιά μου ο πείρα να βοηθήσει να προκύψουν ενδιαφέροντα σημεία εάν ε, έχει χαλαρώσει η σχέση και ορισμένοι θεωρούν ότι όλα είναι δεδομένα δεν ξέρω αν όλα αυτά θα μπορέσω να τα συνοψίσω σε τροπολογίες. Είναι πολύ πιο εύκολο να τα σχολιάζει κανείς από ότι να τα γράψει σε ένα κομμάτι χαρτί. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να επέμβει, τότε θα επανέλθω στην ΚΕΙ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις σας. Δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις γιατί ήμουν σκιώδη στις προηγούμενες εκθέσεις πρωτοβουλίας και έχουμε μια εμπειρία στον διάλογο αυτό τον διευρυμένο. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά καινούρια στοιχεία. Πρέπει να πω επίσης ότι υπάρχει πλήρη στήριξη ε, σχετικά με το ότι οι επιτροπές λογιστικού ελέγχου δεν είναι ανεπίσημα σώματα και πρέπει να έχουν πλήρως μορφοποιημένους τρόπους ελέγχου. Είναι ε, σαφώς ε, επιτροπές οι οποίες ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ε, τυποποιημένα συστήματα λειτουργίας τα οποία να εγκρίνονται από τους μετόχους τους σε αιτήσια βάση και να καλύπτουν όλα τα θέματα όπως και τους διαγωνισμούς και τους λογιστικούς ελέγχους και τις εναλλαγές λογιστικούς ελέγχων και αυτό θα πρέπει να ισχύσει σε μεγάλες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη και εγώ μίλησα όχι μόνο σε βρετανικές εταιρείες αλλά σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Πολλές ε, επιχειρήσεις μεγάλες με διαβεβαίωσαν ότι έχουν αυτά τα μορφοποιημένα πλήρως συστήματα και ε, είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Πιστεύουν ότι αν τυχόν ο παροχέας του λογιστικού έλεγχου, αν παρέχει ε, και ε, άλλες υπηρεσίες εκτός από τον αυστηρά λογιστικό έλεγχο θα πρέπει να αδειοδοτηθεί γι' αυτό από την Επιτροπή ε, Λογιστικού Ελέγχου που υπάρχει στην επιχείρηση. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και εγώ έχω εμπειρία στον τομέα αυτό και με τον τρόπο με τον οποίο πληρώνονται οι λογιστικές υπηρεσίες μέχρι πριν μερικά χρόνια ε, τα λογιστικά των επιχειρήσεων ήταν πάρα πολύ σκοτεινά, στεγανά θα έλεγα. Αλλά μετά το 2008 ο ρόλος του λογιστικού ελέγχου έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Επιχειρήσεις που δεν είχαν επιτροπές λογιστικού ελέγχου τώρα πλέον έχουν. Αυτό έχει βελτιώσει την διαχείριση των επιχειρήσεων και έχει σίγουρα βελτιώσει την άσκηση του λογιστικού ελέγχου τελικά η διαδικασία του ελέγχου, του λογιστικού, είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει κυρίως τους μετόχους και τους ιδιοκτήτες της εταιρείας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σαφές νόμιμο, θα έλεγα, πλαίσιο μέσα στο οποίο να λειτουργεί η επιχείρηση και να ασκείται και ο, ο λογιστικός έλεγχος. Είδαμε επίσης σχετικά με την επιμέρους εναλλαγές ε, λογιστικού, υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου. Εδώ υπάρχει θα έλεγα κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και εδώ θα έλεγα εφόσον υπάρχει εναλλαγή η εναλλαγή θα πρέπει να αφορά το σύνολο του λογιστικού ελέγχου και όχι μόνο επιμέρους λογιστικές ελεγκτικές δραστηριότητες. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει θα έλεγα δραστηριότητες της επιχείρησης που δεν υφίστανται πλήρως τον έλεγχο τον λογιστικό όπως θα έπρεπε. Νομίζω ότι αυτή είναι η συνένεση στην οποία μπορούμε να καταλήξουμε. Όλοι θέλουμε μια ανταγωνιστική αγορά λογιστικού ελέγχου. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε εκεί και ποια μέτρα είναι απαραίτητα και αναλογικά. Δεν θα πρέπει οι επιχειρήσεις, οι ίδιες επιχειρήσεις ή παρόμοιες να δίδουν διαφορετικές απαντήσεις και θα πρέπει επίσης η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου της Επιχείρησης να έχει τα μέσα, τις αρμοδιότητες και τη δυνατότητα να αποφασίζει και να ενημερώνει τους ε, μετόχους. Ε, οι επιχειρήσεις λογιστικού ελέγχου και οι μεγάλες επιχειρήσεις από τη φύση τους και οι μεν και οι δε είναι ε, θα έλεγα επιχειρήσεις παγκοσμίου επίπεδου, σφαιρικού επίπεδου και γι' αυτό τι τη διάσταση δεν θα πρέπει να την αγνοούμε. Υπάρχουν επίση στα πλαίσια αυτών των ρυθμίσεων. you can have no with your Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ρυθμίσει, οι οποίες είναι σε λειτουργία αυτή τη στιγμή που πολύ δεν μου αρέσουν, αλλά αν αλλάζει τους ελεγκτέ σου πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορείς να διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συντοξιοδοτικά προγράμματα των υπαλλήλων σου σαν παράδειγμα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα σχετικά με την πάρα πολύ συχνή εναλλαγή των υπηρεσιών που ασκούν, των εταιριών που ασκούν έλεγχο. Πρέπει λοιπόν τις ρήτρες λέει, να τις εφαρμόσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίσουμε το ενδιαφέρον για αυτές τις ρήτρε και για τους κανόνες τους οποίους αφορούν από πλευρά των επιχειρήσεων ε, εκτός από ένα βέβαια πάρα πολύ μικρό κομμάτι των ρυθμίσεων αυτών που δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμοι. Εγώ προσπάθησα να δω ποιες είναι αυτές οι διαφορετικές οντότητες και εταιρείε στο σύνολο της Ευρώπης. Η ΕΣΜΑ λέει ότι δεν θα πρέπει σαν παράδειγμα να ασκούνται επιπλέον δραστηριότητες, δεν μπορεί να ασκήσει λογιστικές δραστηριότητες. Η EBA μπορεί να είναι καλύτερος χώρος για να ασκήσει αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Εδώ δεν έχουμε αποφασίσει πλήρως ποια από τις εποπτικές αρχές είναι η πιο αρμόδια θα έλεγα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε εμείς ε, να δούμε ε, ποια θα είναι η καλύτερη λύση. Δεν υπάρχει ούτε καν ένας ολόκληρος υπάλληλος στο εσωτερικό της ΕΣΜΑ που να ασχολείται με το θέμα αυτό στις 27 χώρες, που να ασχολείται αποκλειστικά με αυτό. Αυτό είναι γελίο τώρα, είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί ένας υπάλληλος από την ΕΣΜΑ να ασχολείται με τις ρυθμιστικές αρχές από πλευράς ε, των κρατών μελών. Ενώ η EBA βρίσκεται σε ένα ανώτερο επίπεδο και μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των στάνταρτ των επιπέδων που θα πρέπει να γίνονται σεβαστά σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κάποια συνένεση στα σημαντικά θέματα, να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό, να βελτιώσουμε την ποιότητα των ε, ελεγκτικών διαδικασιών αλλά και των μη ελεγκτικών παρεχωμένων υπηρεσιών θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση για να το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 21 Οκτωβρίου, 19 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου. Επί της ουσίας Επιτροπή η νομική θα ψηφίσει στις 18 Δεκεμβρίου. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο, αριθμό 6, που είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2011. Η συγκίτρια είναι η Μαρίσα Ματίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ σε μια σύντομη παρουσίαση της ε, εκθεσής μας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, θα την έχετε κοιτάξει κι εσείς. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τη λογική των προτάσεων αυτών. Όπως γνωρίζετε, προσπάθησα να χωρίσω σε τέσσερα τμήματα το, την έκθεση αυτή, σε τέσσερις βασικούς τομείς. Όχι μόνο όσον αφορά το 2011 και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και όσον αφορά άλλα ζητήματα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής που έχουν να κάνουν με την έκθεση αυτή. Ένα πρώτο τμήμα ασχολείται με την νομισματική πολιτική, ένα δεύτερο με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, το τρίτο αναφέρεται στην Τραπεζική Ένωση και τέλος αναφέρω και μερικά θεσμικά ζητήματα που πιστεύω ότι είναι σημαντικά για την αξιολόγηση αυτή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το πρώτο για την νομισματική πολιτική μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εντοπίσει χαρακτηριστικά στη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2011 που έχουν να κάνουν με την σταθερότητα των τιμών, των πληθωρισμών όπως τα ακούσαμε και από τον ίδιο τον πρόεδρό της στην Επιτροπή μας. Αύξηση των επιτοκίων δυσανάλογα σε σχέση με τον πληθωρισμό μια που οι αξίες αυτές είναι συγκυριακές και όχι διερθρωτικές. Η δεύτερη περίοδος χαρακτηρίστηκε από μια προσπάθεια διόρθρωσης των λαθών που είχαν γίνει κατά το πρώτο στάδιο, με μείωση δηλαδή των επιτεκείων στα τέλη της χρονιάς. Θα ήθελα να κάνω όμως μερικά σχόλια εδώ και να σας αναφέρω τρία παραπάνω σημείο όσον αφορά το 2011. Υπάρχει κάτι ανησυχητικό εδώ που είναι οι επιχειρήσεις και οι οικογένειες τα νοικοκυριά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι τα επίπεδα ρευστότητας που έχουμε στο δεύτερο εξάμενο του 2011 που είναι επίσης κάτι ανησυχητικό διότι μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα μια παγίδα. Τέλος, κάτι άλλο που θέλω εδώ να υπογραμμίσω, έχει να κάνει με την θέση που να μένει είναι σωστή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή ε, διαθεσιμότητα για βοήθεια λόγω της κρίσης, αλλά η τράπεζα αυτή συνέχισε να εφαρμόσει την πολιτική της χωρίς όμως ε, συγκεκριμένες προϋποθέσεις. με αύξηση πιστώσεων ε, στις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις ή αποταμιευτές. Τελικά δεν ήταν αποτελεσματικές οι πολιτικές αυτές. Αυτές είναι λοιπόν οι πτυχές που είχα να αναφέρω όσον αφορά την νομισματική πολιτική. Για το δεύτερο κεφάλαιο, για την οικονομική κρίση, εδώ πρέπει να δούμε τι δουλειά έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια αυτής της κρίσης. Είχε πολιτικές ε, λιτότητας και οι πολιτικές αυτές λιτότητας που εφαρμόστηκαν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες οδηγούν χωρίς αμφιβολία σε ε, την ίδια κατάσταση και στις ε, γύρω χώρες και στις γύρω περιοχές. Είναι κολλητικό κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέτουμε τα εξή ζητήματα. Πρώτον, εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε συζητήσει για την εντολή αυτή. Υπάρχουν προτάσεις για να δούμε κατά πόσο όντω είναι ορθή η εντολή αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή όχι και να δούμε τι μπορεί να κάνει για τον πληθωρισμό και τι συνέπειες μπορεί να έχουν αυτά στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Νομίζω ότι οι συνέπειες αυτές είναι κατάφορες από τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ. Μια δεύτερη ιδέα στο σημείο αυτό έχει να κάνει με το εξή. Ενώ η εντολή της τράπεζας είναι σύντομη, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στην περίοδο αυτής ε, κρίσης ξεπεράστηκε η εντολή αυτή πολλές φορές βάσει του επιχειρήματος που λέει ότι όλα όσα έκανε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και κάνει τα κάνει βάσει επίσημης εντολής. Ήταν τελικά ένας παράγοντας που πάντα συμμετείχε στις συστάσεις και στις αποφάσεις που λαμβάνονται, τις δημοσιονομικές και άλλες, απέναντι στις χώρες μέλη. Ιδιωτικοποιήσεις, δημοσιονομικά, φορολογικά κλπ. Χωρίς αναθεώρηση της συνθήκης ξέρω ότι δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο και να αντιμετωπίσουμε τις ανισορροπίες που έχουμε στην Ευρωζώνη. Αντίθετα, τα προβλήματα συσσωρεύονται. Εκτός αν αποφασίσουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε από τις ρίζες την κατάσταση, να αλλάξουμε ρότα δηλαδή. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να έχουμε μια αλλαγή ρότας. Για τα τελευταία δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, την Τραπεζική Ένωση. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ετοιμάζει την Τραπεζική Ένωση. Πέρα όμως από όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τραπεζική Ένωση υπάρχει και κάτι άλλο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και είναι το εξή. Αν θέλουμε να είναι αποτελεσματική η τραπεζική αυτή ένωση, πρέπει να αποφύγουμε αντιφάσεις. Αντιφάσεις που σήμερα έχουμε μπροστά μας. Για παράδειγμα, η πρόταση αυτή που θέλει να συνδυάσει τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής με συστήματα επίλυσης κρίσεων που να βασίζονται σε εθνικούς μηχανισμούς. Αυτή είναι μια αντίφαση που πρέπει να ξεπεράσουμε. Αλλιώς δεν έχουμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο. Όπως έχω πει και άλλες φορές, πρέπει να προσέξουμε όλος ιδιαίτερος και όλα αυτά που οδηγούν σε ένα κενό ευθύνης όσον αφορά αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και να βοηθήσουν τους πολίτες αλλά να εμπίπτουν μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Αντίθετα, διαπιστώνουμε ότι λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες ε, μερικές φορές δεν συνάδουν απόλυτα με τις δημοκρατικές αρχές. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν την υπερβολή καινού ευθύνη και να δούμε τι ρόλο μπορεί να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, εποπτική αρχή και ως παράγοντα συναπόφασης. Τέλος, για τα θεσμικά ζητήματα που είναι το τελευταίο τμήμα της έκθεσής μου, έχω να σας πω τα Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της που να λάβει υπόψη όλες τις δραστηριότητές της και όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Να δει τι έχει κάνει για τα προγράμματα εξυγίανσης διαφόρων χωρών της Ευρωζώνης. Τέλος, και χωρίς να είναι αυτό λιγότερο σημαντικό, να φροντίσουμε να υπάρξουν γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δεν υπάρχουν ε, σήμερα και πράγμα το οποίο δείχνει ότι δεν τηρείται η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων σε αυτά τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ένα σαφές πρόβλημα και μια αντίφαση με τα όσα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λέει ότι θέλει να αναθέσει υψηλές ευθύνες στον οικονομικό τομέα στις γυναίκες. Αυτά είχα να πω εγώ, δεν ξέρω αν εσείς έχετε να προσθέσετε κάτι, να μας κάνετε κάποιο σχόλιο, να προσθέσετε ιδέες. Αυτό ήταν μια πρώτη συζήτηση και είμαι έτοιμη να ακούσω τα δικά σας σχόλια. Θα τα σημειώσω, θα τα λάβω υπόψη μου. Γιατί πρέπει να δούμε και πάλι το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λαμβάνοντας ε, υπόψη το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον, ε, την ε, εισηγήτρια για τα θέματα που έφυξε και τα τέσσερα θέματα κλειδιά στην έκθεση. Γενικές παρατηρήσεις καταρχήν. Νομίζω ότι είναι μια περιγραφική έκθεση, δηλαδή δεν ε, εστιάζεται σε προτάσεις, δεν, δίνει, δεν προσφέρει κίνητρα και έχει αλλάξει ε, εντολή της ε, τράπεζας από την ε, αρχή. Καταρχήν ε, λοιπόν λέχθη ότι δύο φορές έχει κρίνει και καταδικάσει. Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε γιατί αυτό είναι αιτιολογημένο και γιατί δύο φορές ε, αυξήθηκαν και μειώθηκαν τα επιτόκια. Υπάρχουν ε, ε, αναλύσεις της τραπέζης που εξηγούν γιατί συνέβησαν αυτά και βάσει αυτών διατυπώνονται και οι συστάσεις μειώνεται ε, ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα. Πώς θα λύσουμε λοιπόν μακροπρόθεσμα το θέμα της κρίσεως, πώς θα μπορέσει η τράπεζα να εξασφαλίσει σταθερότητα των τιμών. Τι είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε να αναρωτηθούμε δηλαδή γιατί γίνεται κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τα χρέη των κρατών. Μιλάμε ε, για τις κινήσεις των ε, χρεών των κρατών γιατί αυξάνονται ή μειώνονται και τέλος ε, η γενική μου εξήγηση είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τον πληθωρισμό αλλά και τις θέσεις εργασίας. Είναι θέματα τα οποία ε, επίσης έπρεπε να περιλαμβάνονται στα θέματα που αποσχολούν την Κεντρική Τράπεζα αλλά θα ήταν ε, πιο έγκυρα αν είχαμε μια κοινωνική προσέγγιση η οποία δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνομαι την τοποθέτηση της ηγητρίας διότι ε, η ομοφωνία είναι ε, υπερβολική εφόσον ε, ε, ρυθμίζεται το όλο θέμα από τις συνθήκες που έχουν κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη και άρα είναι ένας νόμιμος θεσμός όσον αφορά την νομισματική πολιτική. Ο εισηγητής λέγει ότι η αύξηση της, ε, του πληθωρισμού το 2009 οδήγησε σε αύξηση των ενεργειακών τιμών όντως αλλά εάν υπάρχει ε, μία διασύνδεση μεταξύ του πληθωρισμού και των ενεργειακών τιμών τότε τι θα γίνει ε, πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση τώρα που υπάρχει στασιμότης και αύξηση τιμών. Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένες υπερβολές τις οποίες θα επιλύσω διμερός με την εισηγήτρια. Στο σημείο 14 ε, μιλάει για την αδράνεια της ε, τραπέζης. Ε, δεν ε, είναι θέμα της ε, ΕΚΤ να αντιμετωπίζει τα χρέη. Υπάρχουν έλεγχοι της ΕΚΤ στα προγράμματα των χρεογράφων και αυτό αναφέρεται στην υπερβολική ρευστότητα. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, την Ένωση των Τραπεζών, ε, είναι ένα θέμα το οποίο ήδη έχουμε καλύψει και έχουμε εξετάσει τις λεπτομέρειες του συστήματος αυτό. Θα το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιαστεί αυτή η έκθεση σε αυτό το αντικείμενο. Όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς, Νομίζω ότι πολύ σωστά οι τράπεζες πρέπει να δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, οπότε χρειάζεται εθνική εποπτεία και εθνικός μηχανισμός ε, χρηματοδότησης. Να διατηρηθεί δηλαδή η εθνική πτυχή σε αυτό το νέο σύστημα της ε, ε, εποπτείας που έχει καταρτιστεί γιατί η ΕΚΤ δεν είναι σε θέση να έχει μία συνολική επισκόπηση των 27 συστημάτων χωρίς να γνωρίζει τις συνθήκες της αγοράς και ε, τις εποπτικές αρχές. Τέλος, ε, ζητάω ο εισηγητής να υπάρξει ε, αυτοέλεγχος ενώ εδώ μιλάμε για ηθική ηθική κατακραυγή. Ενώ αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μία ανάλυση των επιπτώσεων που θα ήταν πολύ πιο χρήσιμες από την αυτοκριτική πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να θέσουμε την ε, τράπεζα υπό τον ε, έλεγχο της της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ίσως χρειάζεται εδώ ένα νέο στοιχείο. διότι οι κανόνες έχουν αλλάξει όσον αφορά την ε, ΕΚΤ και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη Γραμματεία και ίσως στο μέλλον θα πρέπει να καταρτήσουμε μία έκθεση που δεν θα είναι μία συγκεκριμένη ανάλυση της καταστάσεως αλλά θα είναι μία ευρύτερη έκθεση η οποία θα εξετάζει πώς μπορεί να εκπληρωθεί η εντολή της ΕΚΤ και πώς μπορούμε τέλος να κατανοήσουμε ποιος είναι ο στόχος και ο λόγος υπάρξεως της ΕΚΤ. Όσον αφορά τον Πρόεδρο, ο, το, ο έλεγχος της εντολής του είναι κάτι το οποίο κάνουμε συχνά αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετά επικοδομητικός αυτή τη στιγμή διότι οι προτάσεις δεν, είναι, δεν έχουν συνοχή και καλό θα ήταν να γίνει μία έκθεση η οποία είναι πολύ μεστή αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ένα τελικό κεφάλαιο όπως γίνεται σε όλες τις ε, εκθέσεις που θα αναφέρεται στα μιλοντικά χρόνια ή στις ε, αλλαγές και στα ε, τα νέα γεγονότα τα οποία μπορούμε να περιμένουμε. διότι τώρα κάνουμε εκ των υστέρων απλούστατα ε, μία, ε, μία επισκόπηση χωρίς να προσβλέπουμε προς το μέλλον και το τι μπορεί να συμβεί. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα που ήθελα να παρουσιάσω. Ε, θα περιληφθούν και εις, την, τις τροπολογίες μου και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία με το νησηγητή. Ο κύριος Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήλεγξα πολύ προσεκτικά την έκθεση της Μαρίζα Ματία σχετικά με τη δράση της ΕΚΤ το 2011 και συμφωνώ σε πολλά θέματα με τη διάγνωσή της. Ο η συγγήτρια αναφέρεται στις ασυνέπειες της πολιτικής, νομισματικής πολιτικής του 2011 και του αμφισβητήσιμου αποτελέσματος της αυξήσεως των επιτοκίων το πρώτο εξάμεινο του 2011 το οποίο ενέπνιξε ε, μία ντροπαλή ε, αύξηση της ανάπτυξης ε, ενώ το δεύτερο ήμιση του χρόνου ήταν πιο δελακτική ε, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπήρξαν τόσο καλά αποτελέσματα. Η πολιτική μου ομάδα έχει διαπιστώσει ορισμένες αντιφάσεις τις οποίες ανέφερε ο εισηγητής στη δράση της Κεντρικής Τράπεζας και μία ε, αντίφαση ε, για ε, τις ε, απαιτήσει από τα κράτη και όχι από τις τράπεζες. Όταν κοιτά την κατάσταση το, της Ευρωζώνης σε σχέση με τα τεράστια κέρδη της τραπέζης. Όταν λέγεται ότι ο, ο, το, η ΕΚΤ ε, ε, υπαγορεύει τις απόψεις της στα κράτη-μέλη εκεί που δεν της πέφτει λόγος. Τέλος, σε μία ζώνη ευρώ όπου υπάρχουν μεγάλες μακροοικονομικές διαφορές ε, ε, βλέπουμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί η διακυβέρνηση και τέλος να υπάρξει ένα αποτελεσματικό μείγμα πολιτικής, νομισματικής και ε, δημοσιονομικής σε όλα τα κράτη-μέλη διότι ε, ε, εάν κατάφερε να η τράπεζα να υπάρξει ένα χαμηλό επίπεδο επιτοχίων υπάρχει ασθενής ζήτηση υποϊστώσεων και αυτό οδηγεί σε μία έλλειψη επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αναρωτηθούμε αν υπό αυτά σε συνθήκες μπορούμε να ζήσουμε χωρίς δημοσιονομική πολιτική τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και ευρύτερα και αυτό είναι το θέμα που έχει θυγεί σε πολλές εκθέσεις. Εξού και θέλω να συμβάλλω στην ε, ε, έκθεση αυτή και γι' αυτό ε, θα διατυπώσω προτάσεις εν ονόματι της Σοσιαλιστικής Ομάδας για να συμπληρώσω τον κατάλογο του εισηγητή. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα σχόλια για την έκθεση Ματίας. I Θα συμφωνήσουμε σε ορισμένα σημεία όταν μιλάμε για την νομισματική πολιτική. Θα συμφωνήσω μαζί της ότι υπάρχουν προβλήματα με την δυνατότητα δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ορισμένες χώρες στα πλαίσια των, δύο, των ρυθμίσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την οικονομική του στήριξη, τα LTROs. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε. Γιατί είναι προϋπόθεση του να ξεπεράσουμε, για να ξεπεράσουμε την κρίση να αποκαταστήσουμε την χρηματοδοτική ροή προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την κυρία Ματίας. Διαφωνούμε επίσης και για την Τραπεζική Ένωση, αυτά τα οποία λέτε. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες επιπλέον απόψεις που τις οποίες πρεσβεύουμε εμείς, αλλά αυτά που λέτε για την Τραπεζική Ένωση δεν είναι λάθος και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Ανησυχούμε βέβαια και για το θέμα της παρασίας των γυναικών στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει να βελτιωθεί ποσοτικά η παρουσία των γυναικών. Πάντως όταν μιλάμε για την λιτότητα δεν θα συμφωνήσω μαζί σας με αυτά τα οποία λέτε για τη λιτότητα. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, την Ισπανία, με ένα έλλειμμα 9% τέταρτη χρονιά που το έλλειμμα θα είναι ανάμεσα στο 8 και στο 10 και ε, λιτότητα ακόμα δεν έχει υπάρξει λοιπόν στην Ισπανία. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την εισηγήτρια γύρω από αυτό βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν άποψη της σοσιαλιστικής ομάδας θα είναι η ίδια με τις θέσεις ε, ε, της εισηγήτριας. Όταν ήρθε τον προηγούμενο Μάρτιο ο κύριος Σούλτσου στη Βαρκελόνη, έγινε μια συζήτηση μαζί του. και ζητήσαμε και την άποψή του για τα θέματα της λιτότητας και δημοσίου ελλείμματος και είπε ότι είναι υπέρ ενός εξισορροπημένου προϋπολογισμού για να διασφαλιστούν οι παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες μακροπρόθεσμα. Συνεπώς λοιπόν αυτά είναι θέματα θα τα συζητήσουμε εκ νέου. Συναντήθηκε και με τον Γκόραν Πάρσον, τον θέος πρωθυπουργό της Σουηδίας. is, ε, ε, Είναι πρόεδρος ε, μιας Επιτροπής Ανάλυσης της Δασοκομικής Πολιτικής στην Ευρώπη και μας είπε πως αντιμετώπισε τη Σουηδική κρίση το 1994. Κατέβασε το έλλειμμα μέσα σε ένα χρόνο κατά 10% του ΑΕΠ. Αυτή ήταν πραγματική λιτότητα. Και μετά από δύο χρόνια η Σουηδία ξεκίνησε στον δρόμο της λιτότητας. Δεν ξέρω αν θα, ακολουθήσει αυτή την άποψη η πολιτική σας ομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι θέματα τα οποία, στα οποία θα επανέλθουμε. λέτε ότι η λιτότητα είναι βασική αιτία της σημερινής κατάστασης. Κοιτάξτε, ε, οι κακοί πολιτικοί έχουν ε, βρεθεί στα θεμέλια, βρίσκονται στα θεμέλια και προκάλεσαν αυτή την κρίση. Αυτό δείχνουν οι στατιστικές πάντως. Τα προβλήματα είναι σοβαρά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζη δεν είναι υπεύθυνη για την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι σε ορισμένες χώρες της Ένωσης σήμερα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, εμείς θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες γιατί δεν συμφωνούμε πλήρως με τον τρόπο με τον οποίο η εισηγήτρια περιγράφει την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην παρούσα κρίση. Αυτά. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τις τροπολογίες μας και θα συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ε, θα αντικαταστήσει κάποιος τον Σβέν από τους πράσινους. Όχι. Καλώς. Α, Ξέχασα τον Ντέρκ. Α, είναι εδώ η κυρία Εύα Ζολή. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Μαρίζα Ματίας, για την πρώτη της έκθεση. Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε μαζί της για να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση αποδεκτή από την πλειοψηφία. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε λοιπόν την έκθεση με μία σειρά θα έλεγα στοιχείων που θα αφορούν και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2011 αλλά και κάποιες ε, προβλέψεις για την ευρωπαϊκή, την ενισχυμένη ευρωπαϊκή και οικονομική Ένωση. Σε επίπεδο αναδρομικό θα έλεγα θα επανέλθουμε στις αναλύσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στις δύσκολες στιγμές του 2011 στον τομέα της νομισματικής πολιτικής και ιδιαίτερα στην πρώτη προσπάθεια αναχρηματοδότησης από το Δεκέμβριο του 2011 και που απέτρεψε ένα μαζικό credit crunch, λέει στα αγγλικά η ομιλήτρια. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψη της εισηγήτριας στην παράγραφο 6 της ε, πρότασής της. Αυτό που έχει σημασία είναι να εμείνουμε στην απουσία της αιρεσιμότητας για τη χρηματοδότηση ε, και όχι την αντικατάστασή τους από επιδοτήσεις μεγάλου εύρος. Νομίζω ότι υπάρχουν παραδείγματα στην Τράπεζα της Ιρλανδίας σαν παράδειγμα σε συνεργασία με την κυβέρνηση υπήρξαν κάποιες δυνατότητες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ενδιαφέροντα τρόπο. Ένα άλλο σημαντικό σημείο του 11 ήταν η συμμετοχή της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Τρόικα των χωρών που βιώνουν ένα πρόγραμμα ενίσχυσης. Νομίζουμε ότι αυτή η εμπλοκή μπορεί να δημιουργεί κάποιες συγκρούσεις συμφερόντων και θα πρέπει αυτές τις συγκρούσεις να τις προλάβουμε. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Στα πλαίσια λοιπόν της προσπάθειας συνέχειας με τις δύο τελευταίες εκθέσεις, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ζητήσουμε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στην ΕΚΤΑΦ, ιδιαίτερα σε σχέση με τις κατεπίγουσες δυνατότητες ε, ρευστότητας που έχουν οι εθνικές τράπεζες που είναι στο ευρωπαϊκό της Ευρωζώνης και μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να ζητήσουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια για τη σύνθεση του προπολογισμού της ΕΚΤΑΦ ιδιαίτερα στους μη ανταλλάξιμους τίτλους που ανήκουν στο ενεργητικό του Ιδρύματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο ζητάμε εδώ και καιρό, όπως επίσης και τη δημοσίευση των πρακτικών του, του Συμβουλίου Διακυβέρνησης της Τράπεζας. Θα πρέπει επίσης να βρούμε και κάποιες ε, επιπλέον, να καταλήξουμε σε ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον της ενισχυμένης ε, Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης και τι αυτό σημαίνει σε επίπεδο αύξησης του δημοκρατικού ελέγχου. Εξ ονόματος των Πασίνων λοιπόν θα συνεισφέρουμε και εμείς ε, με τις τροπολογίες μας ε, στην έκθεση της κυρίας Ματίας. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι η δράση της ε, τράπεζας ε, της Μεγάλης Βρετανίας με το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι προσπαθεί να κάνει κάτι ίδιο όπως η οδηγία για την ε, ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Αν δεν πετύχει, δεν ξέρω. Είναι δηλαδή μια αντίστοιχη πρόταση. Εμείς θα έπρεπε να πετύχουμε, αν μη τι άλλο. Συνεπώς, πρέπει να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Δίρκ, ευχαριστώ εγώ δεν θα μιλήσω για την Τράπεζα της Αγγλίας. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω την κυρία Ματίας για το σχέδιο εκθεσής της και να πω ότι η πρόσβαση στην ε, ρευστότητα το 2011 ήταν μεγάλη. Επίσης ότι τα LTROs, η μακροχρόνια αναχρηματοδότηση, επίσης βοηθάει για τον δανεισμό στα νοικοκυριά και στις ε, επιχειρήσεις. Η τράπεζα υπολόγιζε 2-3 χρόνια, τελικά ήταν παραπάνω. Πάντως διαφωνώ με άλλες προτάσεις που κάνει η συγγήτρια ιδιαίτερα όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Ενώ είναι διαφορετική η στάση της κυρίας από τη δικιά μου, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην ποσότητα. Τώρα υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν οι ελεγκτικές λειτουργίες. Η τράπεζα αυτή είναι βασικός ο πυλώνας πάνω στον οποίο χτίστηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η τράπεζα αυτή πηγαίνει πέρα από την εντολή της αναλαμβάνει και πολιτικό ρόλο ε, ελέγχοντας και χρηματοδοτώντας ε, ε, δημοσιονομικά ελλείμματα. Με κινδύνους ε, βέβαια που αναλαμβάνει και επαναφέρουμε στην έκθεσή μας. Ηθικού κινδύνου. Έπειτα δεν μπορούμε να τονίσουμε ποτέ αρκετά ότι ο σολογισμός της τράπεζας είναι σε δύσκολη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει γίνει μια κακή τράπεζα, κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ δυσάρεστο και πρέπει να σταθούμε επικριτικά απέναντι στην κατάσταση αυτή. Γι' αυτό θα υποβάλω στην έκθεση της κυρίας Ματίας διάφορες τροπολογίες με επικοδομητικό πάντα πνεύμα. Πρόεδρος, καλώς. Τόμας Μαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ματίας για την έκθεσή της, διότι είναι μία ε, έκθεση η οποία μιλάει καθαρά. Νομίζω ότι μιλάει απροκάλυπτα και παρουσιάζει θέσεις στις οποίες έχω πολλές διαφωνίες όσον αφορά την ε, Τραπεζική Ένωση 20 έως 23. Πρέπει να λειτουργήσει αυτή η Τραπεζική Ένωση. Ποιος θα φέρει την ευθύνη. Διότι δεν θέλουμε να διατηρήσουμε στη ζωή τράπεζες που δεν αξίζουν, αλλά να έχουμε ένα σύστημα χρηματοδότησης που θα χρηματοδοτηθεί αυτεπαγγέλτο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το θέμα μας. Ε, τώρα, αυτό το σκιώδες τραπεζικό σύστημα πρέπει να ε, επιληθεί και ε, υπάρχουν 60.000 τράπεζες. Τι προέχει ο αριθμός των τραπεζών ή οι μεγάλες τράπεζες. Μπορεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να έχει μία εποπτεία. Βλέπω οι πύργοι της ΕΚΤ να ανεβαίνουν και να αυξάνονται ε, αλλά πρέπει να υπάρχει, διαφο... πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των διαφόρων καθηκόντων και θα πρέπει να εμπλακούν και οι εθνικοί οργανισμοί όπως η Μπάρφιν ε, διότι νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό θέμα όπου διαφοροποιούμε από την εισηγήτρια. Όσον αφορά τα θεσμικά θέματα δεν συμφωνούμε διότι μία κριτική ε, αυτοαξιολόγηση δεν επαρκεί. Ε, πρέπει να δούμε τι πήγε καλά, πού υπήρχαν θετικά αποτελέσματα και τι πρέπει να τονίσουμε δεν νομίζω ότι όλοι συμφωνούν με τα μέτρα της ΕΚΤ. Παραδείγματος χάρη να πρέπει να υπάρχουν ε, συνεχή κρατικά δάνεια για ε, χώρες οι οποίες ε, δεν ανταποκρίνονται. Δεν, θα πρέπει τα χρήματα να επιστρέφονται. Δεν είναι χρήματα τα οποία πάνε σε μία μαύρη τρύπα. Επίσης υπάρχουν οικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών αλλά συμφωνήσαμε η ευρωπαϊκό εξάμεινο με συντονισμό, συνεργασία και η θέση μας είναι τελείως διαφορετική και η αξιολόγηση εκεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ σημαντική. Και τέλος συμφωνώ και θα πω ότι στο, στη μελλοντική έκθεση, έκθεση για την ΕΚΤ πρέπει να κοιτάμε προς το μέλλον πού πηγαίνει η κατάσταση, πόσο μπορούμε να ε, θεσμοποιήσουμε ορισμένα θέματα, να υπάρχει εργασία και στο μέλλον γιατί η ΕΚΤ έχει ε, πολλά στελέχη που προσβλέπουν στο μέλλον άρα μπορούν ε, στο θέμα του μέλλοντος να μας δώσουν ένα όραμα κάτι το οποίο να συζητήσουμε συγκεκριμένα αν αυτό δηλαδή πρόκειται να γίνει εδώ στην Επιτροπή μας ή ε, αν θα δώσουμε έναυσμα για συζητήσεις τις οποίες ε, ε, χρειαζόμαστε επιγόντως. Ευχαριστώ η Εστρίντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον την εισηγήτρια για την εργασία της, χωρίς όμως να τη συγχαρώ για ορισμένους προσανατολισμούς της εκθέσεώς γιατί πιστεύω ότι συχνά σφάλει και δεν απευθύνει σωστά τις κριτικές της ή τις προτάσεις σας. Δεν θα επισέλθω εδώ σε λεπτομέρειες. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τροπολογίες και θα το πράξουμε. Θέλω όμως να κάνω μία παρατήρηση γιατί στο σημείο 27 ανησυχεί για την ε, έλλειψη γυναικών στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και θεωρεί ότι αυτό είναι έλλειψη ε, ενδιαφέροντος του Συμβουλίου για ισότητα. Αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποτελείται από τους επικεφαλής των εθνικών τραπεζών των κρατών και γι' αυτό ούτε η Ευρώπη ούτε η ΕΚΤ δεν μπορεί να επιλέξει τους διοικητές των εθνικών τραπεζών. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει σε επίπεδο εθνικό. Και άκουσα κυρία Πρόεδρε ότι ίσως θα σας ενδιέφερε να αναλάβετε τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου. Εξαιρετικό νέο, αλλά καλό θα ήταν να ξέρουμε ε, πόσο πρέπει κανείς να είναι διακριτικός τους επόμενους ε, μήνες για να μην λεχθεί ότι χρησιμοποιήσετε τη θέση σας εδώ για να προωθήσετε την υποψηφιότητά σας. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το ξέρετε και από μόνοι σας. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε και άλλα. Πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι ακόμη σχετικά με τις ποσοστώσεις που πρότεινε η κυρία Ρέντινγκ. Η κυρία Ρέντινγκ ποτέ δεν πρότεινε ε, συμβόλαια, στα διοικητικά συμβούλια, στα στέντε των ανωνύμων εταιριών, ε, στα προεδρία τους, αλλά στα εποπτικά συμβούλια, δηλαδή στα Aufsichtsräte ε, και εκεί Εκεί έχουμε ένα διαφορετικό εταιρικό δίκαιο μεταξύ κρατών, μεταξύ χωρών όπως η Γερμανία, οι βόρειες χώρες και άλλες χώρες οι οποίες ακολουθούν το γαλλικό σύστημα ή τον Απολεόνιο κώδικα. Οπότε ε, πρέπει να προσέχουμε και δεν πρέπει ε, να ε, λοξοδρομούμε. Εάν λοιπόν άκουσα την, ε, σωστά από την διερμηνία ε, η συγγήτρια είπε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τον ρόλο της ΕΚΤ. Νομίζω ότι ο ρόλος της ΕΚΤ εδρεώνεται από τα, συνθήκη. Δεν ε, υπάρχει περίπτωση να θίξουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά για να βελτιώσουμε διάφορες προτάσεις και διαπιστώσεις που παραθέτονται σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ η Σιλβή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια, να συμφωνήσω με τον Ραμόν, τον ε, σκιώδη εισηγητή μας που είναι πιο αρμόδιος από μένα. Δύο θέματα εδώ. Πρώτον πρέπει να αναφερθούμε στην Τρόικα και αυτά τα οποία συμβαίνουν στο όνομα της Τρόικα. Πρόκειται για μια βασική καινοτομία, έχει πολύ σημαντικές συνέπειες για ορισμένες χώρες θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό και λέω στην εισηγήτρια ότι θα καταθέσω τροπολογίες επ' αυτού και επί άλλων θυμάτων. Δεύτερον, να την στηρίξω όταν αναφέρεται στην διαφορετική σύνθεση ε, του Συμβουλίου των Κυβερνητών των Τραπεζών και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί το 2011 αποχώρησε η κυρία Γκούντρουν Βέντελ Τούβερελ και έτσι πλέον η σύνθεση του Συμβουλίου αυτού του οργάνου είναι ε, ασύμβατη με τις ισχύουσες ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν όλα αυτά να συνεχίσουν να μένουν στην έκθεση. Λοιπόν, δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Μαρίζα, μπορείς να κλείσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ φυσικά να απαντήσω σε όλα τα σχόλια τα οποία έγιναν. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως όλους όσους πήραν το λόγο. Υπάρχουν τομείς τους οποίους από ό,τι φαίνεται θα συμφωνήσουμε περισσότερο από ό,τι σε άλλους. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να σημειώσουμε πρόοδο εκεί όπου υπάρχει η δυνατότητα. Για την εντολή των τραπεζών σαν παράδειγμα. Εδώ είναι κάτι με το οποίο μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες. Με τις προϋποθέσεις, την ερεσιμότητα. και το θέμα των δανειοδοτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το θέμα των λεγόμενων κακών τραπεζών. Αυτά είναι θέματα τα οποία μένει ακόμα να εξεταστούν. για τις συνέπειες της ανάλυσης αυτής στο μέλλον. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποιες παρατηρήσεις επιμέρους, σαν παράδειγμα τις συνέπειες που έχει η αύξηση των επιτοκίων από το 2011 και μετά. Υπάρχει μία μικρή αναφορά η οποία λέγει ότι είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί χώρου περισσότερο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι κάποιες από τις επιπτώσεις της εμπλοκής της παρέμβασης στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2011 ήταν ακριβώς να, να ξεπεραστούν τα εμπόδια τα οποία ε, θα υπήρχαν στο δρόμο της ανάκαμψης. Πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς τα επιτόκια σε σχέση με τα επιτόκια με τα οποία το ευρώ ε, γενικά κινείται στις διεθνείς αγορές. Για το 18 τώρα, ίσως εδώ να υπάρχει θέμα διατύπωσης, αλλά η ίδια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέγει ότι η προσπάθεια κερδοφορία της είναι κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με την αγορά των τίτλων και με την αγορά των κινητών αξιών. Τώρα, ίσως κάποιες λεπτομέρειες για τις εξελίξεις στον τομέα και την επιρροή των εξελίξεων στον τομέα των τιμολογίων για την ενέργεια. Εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε να αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας αντίθετα με τα επιτόκια. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Υπάρχει στον τομέα της ενέργειας μηχανισμός εποπτείας και υπάρχουν επίσης και πολλαπλές μορφές απαντήσεων από πλευρά των κρατών μελών στην επίλυση της κρίσης. <clears throat> Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε σχέση κάτι με αυτό, με κάτι το ειδικότερο σε σχέση με τις επιπτώσεις των τιμών της ενέργειας. Ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, είναι η αστάθεια των τιμών. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της ανισότητας ανδρών-γυναικών. Το ότι δεν έχει γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν πρέπει να μας παρεμποδίζει να αντοθέτουμε το θέμα σε καθημερινή βάση, όπου σε όποιο φόρουμ αυτό είναι δυνατόν. Ε, σε κάποιες άλλες, για κάποιες άλλες παρατηρήσεις των συναδέλφων υπάρχουν κάποια προβλήματα πράγματι τα οποία αφορούν την ορολογία αν θέλετε. Ε, μελέτη των επιπτώσεων ας πούμε σε ορισμένες περιπτώσεις, λιτότητα, και πως ε, η λιτότητα εκφράζεται σε διάφορες γλώσσες. Εδώ είναι θέμα το οποίο είναι θα έλεγα πολύ ενδιαφέρον. Είναι θέματα ορολογίας όλα αυτά. Στην Ισπανία πάντως ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει ύφεση οικονομική και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει αντικείμενο συζήτησης. Είμαι λοιπόν στην διάθεσή σας για να συζητήσω όλα τα επιμέρους σημεία τα οποία θέσατε και οποιαδήποτε άλλα θα θελήσετε να θέσετε στις επόμενες μέρες. Θα συμφωνήσω ότι πολλές από τις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει, που, τις οποίες προτείνετε, θα πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο έτσι ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα μείνουν ικανοποιημένοι αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να διανύσουμε όσο μεγαλύτερο διάστημα από κοινού γίνεται. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κάτι παραπάνω από κεντρικός. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Τώρα για την Τρόικα, για τους μηχανισμούς ρύθμισης και εκεί έχει δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να μην αγνοήσουμε. Απαιτείται λοιπόν να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτή τη φάση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 25 Οκτωβρίου. Θα εξατωστούν οι τροπολογίες στις 19 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 21 Ιανουαρίου. Το Φεβρουάριο ελπίζουμε να πάει το θέμα στην Ολομέλεια και να ψηφίσουμε εκεί. Τώρα, περνάμε στο σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη, που είναι η ψηφοφορία της έκθεσης για μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Λοιπόν, για να δούμε, έχουν όλοι τους καταλόγους ψηφοφορίας, τις κάρτες σας. Για βάλτε τις κάρτες σας στο μηχάνημα για να ελέγξουμε. Όπως γνωρίζετε, θα μπορούσε να αποδειχτεί περίπλοκη η ψηφοφορία, αλλά ελπίζω να αποδειχτεί απλή. Υπάρχουν βέβαια πολλές τροπολογίες από τις επιτροπές που γνωμοδοτούν. Είναι μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, έχει αιτιολογικές αναφορές, αιτιολογικές σκέψεις, διάφορες παραγράφους και ένα παράρτημα που περιέχει τις λεπτομερείς συστάσεις. Σε μερικές περιπτώσεις συνδυάζονται μάλιστα. Συνεπώς, για παράδειγμα, στην περίπτωση του 3, 4 και 5 των ομάδων, 3, 4, 5 και 6 ομάδων, τις συμβαστικές τροπολογίες δηλαδή, υπάρχουν και αιτιολογικές αναφορές και αιτιολογικές σκέψεις. Σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε πάντως να βρούμε το δρόμο μας. Επίσης υπάρχουν κάποιες ε, προτάσεις αύκο για αποκλειστικές αρμοδιότητες που ψηφίζουμε έτσι και αλλιώς εφόσον η ομάδα συμβαστικών ε, ψηφιστεί. Δεν έχουν ζητηθεί επίσης κατά τμήματα ψηφοφορία. Σε κάποιες περιπτώσεις το κείμενο ΑΦΚΟ είναι προσθήκη στο κείμενο τη εικόν και όχι αντικατάσταση. Επίσης υπάρχουν ε, και κάποια θέματα της Επιτροπής Προϋπολογισμών που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής και είπαμε ότι θα τις εξετάσουμε σαν επρόκειτο για κανόνα 50, για άρθρο 50 μάλλον, επειδή δεν είχαμε καιρό να διαπραγματευτούμε. Οπότε προτείνω όπου τεθεί τέτοιο θέμα να εγκρίνονται αυτόματα μέσα στην ομάδα ε, τροπολογιών όπου εντάσσονται. Θα σας τα λέμε όλα αυτά. Όσο ψηφίσουμε θα τα ξέρετε, φαντάζομαι και από τους συντονιστές σας. Τα έχουμε πάντως ήδη συζητήσει και έχουν συμφωνήσει. Λοιπόν, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία πρώτα με τις κάρτες. Εντάξει. Ψηφίστε, δηλαδή βάλτε τις κάρτες σας και ψηφίστε δοκιμαστικά για να είμαστε σίγουροι ότι άλλος ένας... Α, εντάξει, ψηφίσατε όλοι 38. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς, είμαστε έτοιμοι τώρα να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Το πρώτο είναι η συμβαστική ομάδα 7. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην... αφκο 36. αφκο 36. Υπέρ. Το βρήκατε. Σαν Πολ το βρήκες. Ωραία. Αύκο 36. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 ήτανε. Στο τέλος της σελίδα 3 ήταν η τροπολογία αυτή. Ε, Σίγεται ήταν υπέρ, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην ΑΦΚΟ 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Να δούμε και πώς πάνε τα νούμερα. Ένας παραπάνω ψηφίζει από τους σοσιαλιστές. Ωραία. Ευχαριστώ. Πέρα της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 21 ψήφι υπέρ, 18 κατά. Αύκο 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι 21 υπέρ, 19 κατά νομίζω. Αύκο 42 υπέρ. Τη 41 δεν την ψηφίζουμε. Για κάποιο λόγο ακαλύπτεται από την ομάδα 6. Την ομάδα συμβαστικών τροπολογιών 6. Είναι τελευταία στιγμή αλλαγή. 41 καλύπτεται από το 6. Οπότε τώρα θα ψηφίσουμε τη 42. Συγγνώμη, διακοπή. Νομίζω ότι η ΑΦΚΟ 41 δεν καλύπτεται και πρέπει να την ψηφίσουμε. Υπάρχει εξάλλου στον κατάλογο ψηφοφορίας. Δεν υπάρχει καμία παράγραφος ε, που να λέει το ίδιο πράγμα στο κείμενο, οπότε γιατί να την εξαιρέσουμε. Μαριάν, τι λες εσύ. Η συγκήτρια θα το και θα μας πει. Επιτρέψτε μου, ναι, κύριε Πρόεδρε, καλύπτεται από τις συστάσεις 4-3 για τον αυξανόμενο ρόλο του Κοινοβουλίου, Εθνικών Κοινοβουλίων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για να μην υπάρχουν επικαλύψεις, γι' αυτό νομίζω ότι σωστά η Γραμματεία ε, είπε ότι καλύπτεται από την συμβαστική ομάδα, την ομάδα συμβαστικών τροπολογιών θέλεις να την ψηφίσουμε χωριστά, σε πειράζει αν δυο φορές μπορούμε να ψηφίσουμε και χωριστά, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι στις αιτιολογικές σκέψεις. Εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτι διαφορετικό στο ψήφισμα είναι μια γενική διάταξη που μιλάει για την ανάγκη για δημοκρατική νομιμότητα κτλ. Στις συστάσεις στο παράρτημα υπάρχει κάτι ξεχωριστό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για μένα. Μπορεί να απορριφθεί, μπορεί να εγκριθεί, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί από την ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε, το συμφωνήσαμε αυτό, λέει Πρόεδρος, ψηφίζουμε την ΑΦΚΟ 41. ΑΦΚΟ 41. Υπέρ παρακαλώ. κατά αποχές νομίζω ότι η ίδια πλειοψηφία είναι ότι εγκρίνεται 21-19 αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άλλος ένας πρέπει να ψηφίσει. Εντάξει, εγκρίθηκε 20-18 το αποτέλεσμα. Αύκο 42. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Αύκο 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ομάδες βασικών τροπολογιών 2 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, καλά, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Είπαμε ομάδα συμβαστικών τροπολογιών 2. Εγκρίνεται 28 ψήφι υπέρ, 11 κατά. Και τώρα πάει με απασχόλησης στη σελίδα 12. Σελίδα 12. Απασχόλησης Α. 13 τελικά είναι, σελίδα 13 διορθώνει ο πρόεδρος. Απασχόλησης Α, ε. Το βρήκατε? Στο τέλος, end of block 2 μετά. Λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απασχόλησης Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απασχόληση Σ, Γ, τι έγινε, διαμαρτυρίες από την αίθουσα. Για ψάξτε στη σελίδα 13, θα το βρείτε. Εκεί που λέει end of block 2. Αμέσως μετά. Το βρήκατε. Το βρήκατε, βρήκατε πού είναι. Το βρήκανε. Ωραία. Απασχόλησης C, γάμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόλησης D, δέλτα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόλησης ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται απασχόλησης H ή τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόλησης I τα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε εντάξει δεν σηκώνονται τα χέρια ομολογώ απασχόλησης I λοιπόν Ι ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Άλλος ένας. Πέρα τη οφορίας. Απορρίπτεται 15 υπέρ, 24 κατά. Απασχόληση κάπα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται απασχόληση Έλα. λάμδα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται απασχόληση M υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται απασχόληση ένα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης ο όμικρον υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης P υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης Q υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης R υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, ομάδα συμβαστικών τροπολογιών 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην ΑΦΚΟ 8 που είναι στη σελίδα 25. 25 σελίδα. Στην τελευταία, εκεί που λέει End of Block 3. Το βρήκατε. Αύκο 8 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές. Δεν ε, καταλαβαίνω πώς ψηφίζεται. Εγκρίνεται. Αλλά ας το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε. Αυτό είναι το καλύτερο. Ψηφίστε παρακαλώ. Άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 υπέρ 18 κατά. Απασχόλησης U. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα λοιπόν περνάμε στην τροπολογία 408. 408. Η επόμενη σελίδα δίκη σε βλέπω μπερδεμένη. Τροπολογία 408. Είναι η αρχή του δεύτερου τμήματος, αν το ξεχωριστό ξεχωριστή δέσμη χαρτιών. Έτσι, ωραία. 408, λοιπόν. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 409 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 410 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 411 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ομάδα συμβαστικών τροπολογιών 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη σελίδα 5, εκεί που λέει End of Block 4. Πρόκειται για μια προφορική τροπολογία που έχω υποβάλει εγώ. Θα σας ε, εξηγήσω. Μιλάει για την ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που μου ζητήθηκε να συμπεριλάβω. Η Eurostat το ζήτησε. Η εισηγήτρια συμφώνησε με την τροπολογία αυτή. Διαφωνεί κανείς να την ψηφίσουμε? Όχι, ωραία. Συνεπώς, ψηφίζουμε την προφορική αυτή τροπολογία της Προέδρου αριθμό 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. αποχέ. εγκρίνεται. Προφορική 2 τώρα υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Έρχομαι τώρα της Άλντε, μια προφορική τροπολογία αριθμό 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Προφορική τροπολογία αριθμός 1 της Άλντε. Ψηφίστε παρακαλώ. Που προσθέτει το whereas the European Treasury should be set up κτλ. Το οποίο βέβαια συμπίπτει κάπως με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ψηφίσατε όλοι. Άλλοι δύο. Πέρασε της ψηφοφορίες, Εγκρίνεται 20 υπέρ 18 κατά. Τώρα ερχόμαστε στην δεύτερη προφορική τροπολογία της Άλντε, Common Insurance. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα το λέξω και αυτό γιατί δεν ψηφίζεται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ψηφίστε. Άλλος ένας. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20-20 είναι το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται λοιπόν. Τώρα πάμε. Απασχόληση Β υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση W υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης X υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και απασχόλησης Z υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης AA υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμών C υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΑΦΚΟ 16 υπέρ κατά αποχές. Α, μια στιγμή. Αύκο 16 λέει, αλλά στην πραγματικότητα είναι 17. Ναι, κάποιο email κυκλοφόρησε. Μαριάν, είσαι εντάξει ότι πρόκειται για την ΑΦΚΟ 17 στην πραγματικότητα, εκεί που λέει 16. Στα αριστερά λέει αιτιολογική σκέψη CB, B μικρό, νέο. Αυτό είναι το σωστό. Και εκεί που λέει 16 είναι 17 στην ΑΦΚΟ. CBB, ναι. Που λέει εφόσον το ESM μπορεί να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο μέσω της ρίστρας ελαστικότητας άρθρο 352 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. κλπ. Εντάξει, καταλάβατε τι ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το επόμενο είναι ΑΦΚΟ 18 πάλι τυπογραφικό. Το CBC. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αύκο 19 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αύκο 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε. Αύκο 10. Ψηφίστε παρακαλώ. Δύο ακόμα πρέπει να ψηφίσουν. Ψηφίστε ή αλλιώς κλείνω την ψηφοφορία. Απορρίφθηκε 16 υπέρ, 21 ψήφι κατά, απορρίπτεται. Αύκο 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 αύκο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αύκο 13 υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά να το ελέγξουμε Αύκο 13 λοιπόν ψηφίστε παρακαλώ Ψηφίσατε όλοι άλλος ένας Εντάξει, εγκρίθηκε 21 ψηφί. υπέρ, 20 κατά. Αύκο 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, ομάδα συμβαστικών τροπολογιών 5. Υπέρ παρακαλώ. Α, πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη σελίδα 10, εκεί που λέει End of Block 5, και έχουμε δύο προφορικές τροπολογίες της Προέδρου, η τρία πρώτα, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται, τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης AB, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης AC, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης AF, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης AD υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης AE υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αύκο 22 υπέρ κατά αποχές Σύγχυση. Λοιπόν, αύκο 22. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αύκο 22. Ψηφίστε. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Άλλος Όλο Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 20-20 είναι το αποτέλεσμα. παρακαλώ. 20. Τώρα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ομάδα σεβαστικών τροπολογιών 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε τώρα εκεί που λέει End of Block 6, σελίδα 15, προφορική τροπολογία 5 της Προέδρου, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης AG, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Αύκο 31, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αύκο 32, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Όσοι έχετε ξεχωριστούς καταλόγους πηγαίνετε στο τρίτο πακέτο. Δεν θα πρέπει να ψηφιστεί το τρίτο τμήμα, έτσι και αλλιώς έχει ολοκληρωθεί αυτό. Περνάμε στο τέταρτο τμήμα, συμβιβαστική ε, ομάδα τροπολογιών υπάρχουν τέσσερα Λοιπόν τώρα στα παραρτήματα το πρώτο είναι τμήμα της ομάδας 4, προϋπολογισμός 2 λοιπόν. Κοιτάξτε, παρακολουθήστε με για μία στιγμή. Είμαστε στη σελίδα 4 του τελευταίου τμήματος. Προϋπολογισμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προϋπολογισμός 4 υπέρ. Για μια στιγμή, για μια στιγμή. Στο τέλος της ομάδας 4, προϋπολογισμός 4. Κλείσαμε με τον προϋπολογισμό 2, το ψηφίσαμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κάποια σύγχυση. Ας πάμε λίγο πίσω στον προϋπολογισμό 2 για να ελέγξουμε πλήρως τον προϋπολογισμό 2. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα προϋπολογισμός 4, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απασχόληση 3, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστικό 5 δεν το, ψοφίζ, δεν το ψηφίζουμε γιατί έχει ολοκληρωθεί εκεί. Πάμε στο τέλος της προσθήκης 4 του παραρτήματος μάλλον 4. Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουμε ψηφίσει στην ομάδα 6. Πηγαίνουμε τώρα στην τελευταία σελίδα, τέλος του έκτου τμήματος, προϋπολογισμός 5. Τελευταία σελίδα, προϋπολογισμός 5, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τώρα ψηφίζουμε το τροπολογημένο κείμενο παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ένας ακόμη πρέπει να ψηφίσει. Τέλος της ψηφοφορίας. 32 υπέρ. 7 κατά. Μία αποχή. Συγχαρητήρια. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Διαδικαστικό. Κοιτάξτε, η, η Μάριον πρώτη. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Πρόεδρε, Νομίζω ότι με το αποτέλεσμα αυτό 32 υπέρ 7 κατά και μία αποχή νομίζω ότι στηρίζουμε ευρέω ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και όπου υπάρχουν θέματα τα οποία κατά το παρελθόν μα έχουν διχάσει κατά πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν του και όδης αλλά και όλου του συναδέρφους που συνεργαστήκαμε μαζί. Μαζί κοπιάσαμε πολύ για να επιτευθούν οι συμβιβασμοί και τώρα έχουμε ένα ισχυρό κείμενο το οποίο θα προτείνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ ψηφίζουμε ένα νομοθετικό κείμενο που σημαίνει ότι έχουμε και κείμενο με ερωτήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε από την πλευρά της δουλειά. Οπότε Ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους. Νομίζω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ καλά μαζί και το ότι όλοι προετοιμαστήκαμε να ρίξουμε όλοι λίγο νερό στο κρασί μας βοήθησε πολύ και οδήγησε σε ένα πολύ καλό πακέτο συμβιβαστικών τροπολογιών και τελικά καταλήξαμε να έχουμε μια απλή ε, ψηφοφορία παρόλο που ξεκινήσαμε με πάνω από 900 τροπολογίες. Ευχαριστώ επίσης και τη γραμματεία. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αποφασίσει ότι έπρεπε έγκαιρα να είμαστε έτοιμοι για να προλάβουμε τη διάσκεψη κορυφή της 18 Οκτωβρίου και το καταφέραμε αυτό επειδή πολλοί δούλεψαν μέρα νύχτα Σαββατοκύριακα και ξέρω ότι αυτό το έκαναν και τα άτομα από τη γραμματεία της ΕΚΟΝ, όχι μόνο οι δικοί μου συνεργάτες αλλά και η γραμματεία της Επιτροπής μας. Έτσι καταφέραμε να ψηφίσουμε καλά και γι' αυτό ευχαριστώ από βάθους καρδίας και την γραμματεία της Επιτροπή μας, οι οποίοι φρόντισαν τόσο πολύ για αυτή την ε, κατάληξη. Να έχουμε δηλαδή μια ισχυρή θέση και με αυτήν να πάμε στο Συμβούλιο. Ξέρετε όλοι ότι με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση Είμαστε σε βαθιά κρίση. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου. Γι' αυτό αυτά που ζητάμε εδώ πιστεύω ότι είναι κάτι θετικό και θα μας, στηρίξει, θα μας στηρίξει ο κόσμος, γιατί χωρίς τη στήριξη του κόσμου, χωρίς δημοκρατική βάση, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Είναι και μερικά άλλοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Οι σκιώδεις πριν φτάσω σε ένα Βέρνες, έχω δύο όμως. Τι θέλεις, να προσθέσουμε μια ψήφο δεν λειτουργήσε η, ψη... κάρτα μου ε, για να ψηφίσω και ήθελα να καταψηφίσω. Αυτό θα ήθελα να σημειώσετε διότι δεν λειτουργήσε. Εντάξει, ένας ακόμη κατα... Ε, εναντίον Φιλίπ, ζήτησε και εσύ το λόγο. Είναι διαδικαστικό κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι οι ομάδες αυτές των συμβιβαστικών τροπολογιών είναι σαν τα συσκευασμένα προϊόντα και αυτό είναι το νέο βήμα το νομοθεσίας καινοτόμου με ομάδες ε, τροπολογιών, ομάδες ομάδων τροπολογιών δεν τα κατήρτισα εγώ, Ρομπέρτο και μετά η Σιλβή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Τάισεν και την Πρόεδρό μας για μια εξαιρετική συνεργασία. κανόν 50 δεν είναι πάντα εύκολο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πήγαν όλα καλά. Πρέπει να σας ευχαριστήσω Νομίζω ότι και για τους άλλους ΣΕΡΠΑ μπορώ να πω ότι όλοι θεωρούμε ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα. Έχουμε ένα κείμενο που ψηφίστηκε από πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές και ότι το καταφέραμε αυτό πριν από το Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικό. Σοφή. Σοφή. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που προσπάθησε να συνδυάσει τόσες τροπολογίες μέσα σε μια εβδομάδα δέκα μέρες και πρέπει να σας πω ότι δεν φταίει η συγγήτρια αλλά νομίζω ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι ικανοποιητική. Είχαμε τόσο λίγο χρόνο και τόσες πολλές τροπολογίες για ένα πολύ σημαντικό θέμα που στο τέλος δεν μπορούσαμε να εκφραστούμε επί των σημαντικών πολιτικών θεμάτων και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι δυσάρεστο ότι αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο αργά αποκρίνεται στην κρίση για ένα θέμα που σοβεί εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια με μικρά βήματα και σε μια εβδομάδα πρέπει να διεκπαιρεώσουμε το θέμα αυτό, πράγμα το οποίο δεν μας επιτρέπει να διατυπώσουμε μια ισχυρή πολιτική στάση γιατί δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε διεξοδικά τις βασικές εναλλακτικές μας λύσεις. Η Σαγήτρια έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Ο καθένας υπήρξε όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος αλλά πολύ με λυπεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δυσκολίες με το χρονοδιάγραμμα αυτού του θέματος αλλά έπρεπε κάτι να γίνει πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε ακόμη την Ολομέλεια όπου ενδεχομένως θα μπορέσουμε να προβούμε σε πιο σημαντικές προσθήκες αλλά ίσως καλύτερα είναι να κάνουμε κάτι λίγο παρά τίποτα. Ο πρώτα. Ευχαριστώ. Απλώς Θέλω να ευχαριστήσω την Μάριαν και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την εργασία για το επικοδομητικό και υπεύθυνο κλίμα στο οποίο όλοι εργαστήκαμε. Η Σόφη ε, συζήτησε τις προθεσμίες αλλά έπρεπε να διατυπώσουμε την πιο ισχυρή θέση πριν το Συμβούλιο και θέλω να ευχαριστήσω το ΕΛΚ που μπόρεσε να περιλάβει ένα ε, κοινωνικό σύμφωνο κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Τώρα ο Τόμας Μαν και μετά ο Βέρνερ. Ε, ήθελα καταρχήν να συμφωνήσω με την κυρία Ίνφελτ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι ε, πηδάμε από τη μία διάσκεψη κορυφή στην άλλη και ε, αυτή η κατάσταση μας παρασύρει. Τρέχουμε σαν τους τρελούς και με συγχωρείς. Μαριάν, σε ευχαριστώ και πάλι για την εξαιρετική σου δουλειά παρόλο που υπήρξε μια κατάσταση που κανείς δεν ήξερε πώς ε, αν είχαμε δίκιο ή όχι. Είναι ε, σαν μία ψυχρολουσία και ουσιαστικά δεν έχει τίποτα να κάνει με τη Μαριάννα. Απλούστατα συμπιέζεται το χρονοδιάγραμμα. Οι πολίτες ζητούν συγκεκριμένες ε, απαντήσεις και αποφάσεις και εμείς πρέπει να σκεφτούμε τι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ τη Μαριάν για τη δουλειά της και πιστεύω ότι στο τέλος το αποτέλεσμα μας αφήνει σκεπτικούς και ο Βέρνερ και μετά ο Σβέν. Θα ήθελα να ε, συμφωνήσω με τη συνάδελφο Ίνφελτ διότι όντως ε, το κείμενο υπάρχει μόνο αγγλικά και μας είπαν από την Προεδρία ότι έπρεπε να επιδοθεί ε, πριν από την διάσκεψη κορυφής αλλά και όχι στην Επιτροπή ιδίω όταν δεν μπορούμε να διαβάσουμε το κείμενο στην μητρική μας γλώσσα. Δεν μπορεί να είναι αυτό το σημείο εκκινήσεως. Είναι κυρία κυρίαρχο, το κυρίαρχη Ολομέλεια η οποία θα συνεδριάσει μετά τη διάσκεψη κορυφή. Σα παρακαλώ. Ο Σβέν. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τη Μάριαν Τάισιν για τη δουλειά που έκανε εδώ. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να τονίσουμε. Υπήρξαν πάρα πολλές τροπολογίες και νομίζω τώρα ότι όλα αυτά τα θέματα ήταν τελείως καινούρια. Πρέπει να σας πω ότι εκπλήσωμε γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε επί χρόνια και πολλά έχουν ε, εδρεωθεί, έχουμε δεδομένες ε, ε, θέσεις και γι' αυτό ε, μπορέσαμε να καταλήξουμε τόσο γρήγορα στην ψηφοφορία γιατί αν όλα αυτά ήταν νέα θα ήταν σαν να ξεκίνησε η ευρωπαϊκή κρίση και έπρεπε να ανταποκριθούμε άμεσα αλλά έχουμε κάνει τόσες ψηφοφορίες επί του θέματος της ευρωπαϊκής κρίσεως οπότε ηρεμήστε δημοκρατικά όμως συμφωνώ ότι πρώτα πρέπει να πάει στην Ολομέλη όπως είπε ο Βέρνερ και μετά η Επιτροπή Οικονομικών κοινωνικών είναι ε, και συγκεντρώνει τους ε, ειδικού για οικονομικά θέματα σε συνδυασμό με την ΑΦΚΟ είναι βασικές επιτροπές δίνει ένα σημαντικό μήνυμα και αν δείτε ε, θέματα σημαντικά όπως οι ενώσει τραπεζών φτάνουν στο Συμβούλιο χωρίς συζήτηση από τη μια μέρα στην άλλη με ένα συμβιβαστικό κείμενο τουλάχιστον εμείς αυτή τη στιγμή καταρτήσαμε μία έκθεση και ε, συμβιβαστικές προτάσεις κατά τρόπον ώστε να μην χάσουμε την νομιμοποίηση της εργασίας μας γιατί αν μετά από τόσες εβδομάδες συζητήσεως δεν αποδίδουμε απλώς διαχειριζόμαστε τις κρίσεις και πολλές φορές μας έχει εκτρέψει η πορεία του Συμβουλίου οπότε δεν πρέπει να μειώσουμε την νομιμοποίηση νομιμοποίηση της δουλειάς μας η οποία διαρκεί εβδομάδες συγχαίρω τη Μαριάν και είδα πόσο γρήγορα μπορείς να εργαστείς για να συμβιβάσεις τόσες πολλές τροπολογίες. Οπότε θα προβαίνουμε σε τροπολογίες και θα αφήνουμε μερικές για σένα να ρυθμίσεις. Ο Ζων Πολ τώρα. Καταρχήν θα ήθελα να ε, συγχαρώ την ε, Μαριάν για αυτή την εργασία η οποία της πήρε πάρα πολύ χρόνο όταν λέει για νυχθήμερα και συμφωνώ. Αλλά για πολλά θέματα πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο αργεί πολύ και χάνει την αξιοπιστία του στο Συμβούλιο. Ενώ τώρα μαζί με τη Μαριάν σεβαστήκαμε τις ε, προθεσμίες για να υπάρχει μία μία έκθεση στην Ολομέλεια και συμφωνώ με τον Βέρνερ αλλά θα έχουμε ήδη μία, ένα πρώτο σχέδιο της εκθέσεως πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το θέμα είναι αν είμαστε έγκαιροι επηρεάζουμε ή όχι. Και αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί για να δούμε εάν ε, τρέχοντας, ε, πηγαίνοντας ε, με βήματα χ μπορούμε να επηρεάσουμε την έκβαση ή αν η έκθεση αυτή, το έγγραφο αυτό, όσο καλό και να είναι, θα μείνει κατά μέρος και ε, θα χρειαστεί να γίνει μια πολιτική συζήτηση και δεν θα πρέπει να μας λένε ότι πάντοτε το Κοινοβούλιο χρειάζεται μήνες για να προχωρήσει και πρέπει να εγκαταλείψουμε την κοινοτική μέθοδο τη στιγμή που εσείς δεν λαμβάνετε υπόψη τα θέματα που συζητούνται στο Κοινοβούλιο και γίνεται η εργασία των ε, ε, εκπροσώπων του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και πιστεύω ότι σε αυτό το βασικό ε, φάκελο και αντιλαμβάνομαι και τη θέση ορισμένων ότι δεν είναι ανεκδοτική συζήτηση ή πρέπει να δούμε εάν κινούμαστε και εάν μας ακούει το Συμβούλιο ή όχι αν όχι πρέπει από κοινού να σκεφτούμε ποια είναι τα συμπεράσματα που πρέπει να αποκομίσουμε από αυτή την κατάσταση. Η Μαριάν βεβαίως πρέπει να μιλήσει τελευταία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας. Όμως συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι εδώ ολοκληρώνεται μια δημοκρατική διαδικασία. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και στις διακοπές. Δηλαδή Ακόμα και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ετοιμάσαμε ένα έγγραφο με την γραμματεία της ΕΚΟΝ και όλες τις ερωτήσεις ετοιμάσαμε που θέλαμε να θέσουμε. Οπότε ετοιμάσαμε, προετοιμάσαμε την ακρόαση που θέλαμε να είχαμε. Κατά τη διάρκεια των διακοπών τώρα και περιμένοντας την ακρόαση ετοιμάστηκε ένα σχέδιο έκθεσης και βασιστήκαμε σε όλα όσα είχαμε ψηφίσει νωρίτερα. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα καινούριο πέρα από την Τραπεζική Ένωση, αλλά και εδώ κάποιο κομμάτι μόνο είναι. Οπότε καταλαβαίνω την κριτική σας, αλλά συμφωνήσαμε να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα και να αφήσουμε όλα σε εκκρεμότητα. Από εκεί και πέρα είχαμε τη βάση και η βάση αυτή, όπω σα είπα, ήταν κάτι που είχαμε ήδη ψηφίσει κατά το παρελθόν εδώ, άρα δεν ήταν τίποτα καινούριο. Οπότε καταλαβαίνω του συναδέρφους που θέλανε μια μικρή αποχρωσή εδώ, κάποια προσαρμογή εκεί κτλ. Και τα κάναμε, γιατί ακριβώς μέσα σε μια δημοκρατική διαδικασία αυτό προβλέπεται. Και έτσι σήμερα καταλήγουμε να μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έγινε πολύ σκληρή δουλειά και όσοι θέλανε να διαβάσουν το κείμενο το διαβάσανε, κάνανε τον κόπο και το διαβάσανε. Υπάρχουν πολλοί που το διαβάσανε και πολλοί ήρθανε να μου πούνε εκεί λείπει ένα κόμμα ή εδώ ένα τόνος ή ξέρω εγώ τι. Άρα πολλοί είναι που διαβάσανε λεπτομερώς το κείμενο. Τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα έτσι όπως το προβλέψαμε. Ήταν ο μόνος τρόπος για να καταλήξουμε. Η συζήτηση έγινε από την αρχή για την διαδικασία το κατά πόσο προλαβαίνουμε μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα ή όχι. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο, αποφασίσαμε όμως παρόλα αυτά να το κάνουμε. Και κάναμε αυτό που σας είπα και πριν. Όταν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ακουστεί η φωνή του, φροντίζει και κάνει τα πράγματα έγκαιρα. Ήδη από τον Ιούλιο λοιπόν υπήρχε ένα κείμενο με τους, από τους τέσσερις προέδρους για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το διαβάσαμε αν τώρα κάποιο πει ότι δεν προλάβαινε και δεν το διάβασε και δεν προλάβαινε για τώρα που είμαστε ήδη μέσα Οκτωβρίου, ε, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τη δομή του Κοινοβουλίου τότε. Εγώ είμαι υπέρ του να μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες όλα τα έγγραφα, αλλά μερικές φορές αυτό είναι πραγματικά αδύνατο και τώρα έπρεπε να δώσουμε την προτεραιότητα στο μήνυμα που θέλαμε να στείλουμε. Γι' αυτό ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλου του συναδέλφους και πιστεύω ότι είναι κάτι θετικό και για το Κοινοβούλιο και για του πολίτε. Γιατί οι πολίτε μερικέ φορέ θέλουν να έχουν την αίσθηση ότι εισακούγονται και νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Προέδρο. Ωραία. Ολοκληρώνουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ όλου. Έληξε η συνεδρίαση. Επόμενη συνεδρίαση είναι την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο στις 7 το βράδυ.